Αγαπητοί συνάδελφοι, okay, we can... Uh, μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ας εγκρίνουμε πρώτα την ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, να εγκρίνουμε χωρίς αλλαγές την ημερήσια διάταξη. Πάμε στο σημείο 4 τώρα. Ανακοινώσει του Προέδρου. Θα οργανώσουμε έκτακτη συνεδρίαση στο Στρασβούργο, Δευτέρα 27 Απριλίου, 7 το απόγευμα, για να ψηφίσουμε κατεπηγόντως μία χρονομοδότηση και να έχουμε και ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Αρίες Κανιέτε για την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2015 και τις προτεραιότητες για τις κλιματικές αλλαγές για το 2016. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε κάποιες δυσκολίες στο έργο της Γραμματείας μεταξύ 2 και 12 Απριλίου εξαιτίας των εργασιών που πρέπει να γίνουν για να αφαιρεθεί ο αμύαντος από τα κτίρια στα οποία δουλεύει η γραμματεία. Οπότε θα υπάρξουν προβλήματα 2 με 12, 2 12 Απριλίου. Οι εργασιακές συνθήκες για τα μέλη της γραμματείας θα είναι δύσκολες αντίξωες ε, στην περίοδο αυτή και κατά πάσα πιθανότητα αν δεν ολοκληρωθούν τα έργα φέρει στο αμιάντου να παραταθούν κατά μία εβδομάδα οι δυσκολίες. Οπότε περιμένουμε κάποιες καθυστερήσεις ε, στις ε, απαντήσεις της γραμματείας και θα έχουμε δυσκολία και πρόσβαση στη γραμματεία, ακόμη και τηλεφωνικά. Σε ό,τι αφορά τη διερμηνία, έχουμε διερμηνία σε 21 γλώσσες για την πρωινή συνεδρίαση και 22 το απόγευμα. Το πρωί δεν έχουμε στονικά και μαλτέζικα και το απόγευμα δεν έχουμε στονικά. Έχετε λάβει ηλεκτρονικά από το e-meeting το φάκελο της Επιτροπής και θα γίνει και μετάδοση απευθείας από το διαδίκτυο. Σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης τώρα. Έγκριση των πρακτικών της 17ης Δεκεμβρίου του 2014. Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, τα πρακτικά θα θεωρηθούν ως εγκεκριμένα. Και περνάμε στο κυρίως θέμα την παρουσίαση της κατάστασης και των προοπτικών ε, του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος για το 2015 από τον Διευθυντή της, ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, τον κύριο Μπρένιξ, στον οποίο και θα δώσω πάρα αυτό το λόγο για να μας κάνει την παρουσίαση της έκθεσης για το 2015 ε, και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση. Σα Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε την πενταετή έκθεση για την κατάσταση και την εικόνα ε, του περιβάλλοντος ε, στην Επιτροπή σας. Να σας πω ότι την εβδομάδα που ξεκίνησε η έκθεση, πριν από τρεις εβδομάδες, υπήρξε και μία εκδήλωση την οποία χρηματοδότησαν κάποια από τα μέλη της Επιτροπής, ο κύριος Φαρία, ο κύριος Ζαβόρ και η κυρία Ντάλη. Ε, υπήρξε μεγάλη συμμετοχή και από πλευρά σας και θα πρέπει να σας πω ότι ε, χαίρομαι διότι στην αίθουσα είναι εδώ ο Μάικολ Σκούλες και ο Κρίστιαν Χέις οι οποίοι είναι οι δύο εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχουν διαδραματίσει πολύ επικοδομητικό και πολύ σημαντικό ρόλο ε, στα όσα παρουσιάζουμε εμείς εδώ σήμερα. Κάθε πέντε χρόνια το Ευρωπαϊκό, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος συγκεντρώνει τις καλύτερες γνώσεις που έχει για το περιβάλλον και αυτό γίνεται ε, με τρεις τρόπους. Αναφέρουμε την κατάσταση του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος, το συνδέουμε αυτό με το θεματολόγιο των πολιτικών μας ε, και βλέπουμε πού υπάρχει πρόοδος και πού υπάρχουν κενά και επίσης εξετάζουμε και ε, τι ακριβώς μπορεί να γίνει στο μέλλον και το τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε. Αυτή τη φορά, λόγω της ε, πολιτικής σημασίας της ανάκαμψης από την κρίση, υπάρχει επιπλέον προσοχή σε θέματα καινοτομίας και επενδύσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν προκειμένου προκειμένου να ενισχύσουν το περιβαλλοντικό θεματολόγιο και ταυτόχρονα και το θεματολόγιο για μια πράσινη και γαλάζια οικονομία. Ε, η έκθεση είναι μια σύνοψη η οποία πλέον έχει μεταφραστεί σε 23 γλώσσες. Οι υπόλοιπες γλώσσες ε, θα ακολουθήσουν πολύ σύντομα και το όλο θέμα ε, πλαισιώνεται με βάση τις ε, παγκόσμιες megatrends, ε, διότι το περιβάλλον θα πρέπει να ληφθεί υπόψη με βάση την παγκόσμια διάστασή του. Η έκθεση έχει 25 τετρασέλιδες ενημερώσεις για ε, μια σειρά από περιβαλλοντικά ζητήματα, από την ποιότητα των υδάτων σε θαλάσσια θέματα, σε μετριασμό των ε, ε, συνεπειών του κλίματος, στην πράσινη οικονομία και στην περιβαλλοντική υγεία. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε διαδικτυακά βεβαίως. Για εννέα σημαντικά ζητήματα συγκρίνουμε ε, τις 39 χώρες ε, που αφορά η έκθεση. Έχουμε τις 28 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, συν τον, τις χώρες ΕΖΕΣ και 6 βαλκανικές χώρες και ζητούμε από όλες τις χώρες να μας δώσουν αυτή την τετρασέλιδη ενημέρωση και από εκεί και πέρα υπάρχουν και τρεις περιφερειακές ενημερώσεις οι οποίες αναφέρονται στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα δράσης, τον Εύξηνο Πόντο, τη Μεσόγειο και την Αρκτική στην έκθεση προσπαθούμε να προσδώσουμε κάποια αξία σε τρία χρονικά πλαίσια. Ε, το πρώτο είναι το κοινοτικό κεκτημένο και οι καθημερινές εκθέσεις για την ποιότητα των υδάτων, για την ποιότητα του, ε, του περιβάλλοντος, η βιοποικιλότητα ε, και λαμβάνουμε υπόψη τα στοιχεία αυτά, αλλά επίσης έχουμε κατά νου και το 2020 και το 2030 ως βασικό πλαίσιο για τη χάραξη της πολιτικής μας και κάτι που είναι σημαντικό όχι μόνο για το κλίμα αλλά και για τη βιοποικιλότητα, για την αποδοτικότητα προς τους πόρους, ε, για θέματα που αφορούν τη διαχείριση απορριμμάτων και όπως γνωρίζετε, η Ευρώπη έχει και ένα θεματολόγιο για το 2050 στο 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, το οποίο ε, ε, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μια κυκλική οικονομία που ε, σχετίζεται και με ισχυρή βιοπικιλότητα για προσαρμοστικές κοινωνίες και ανάπτυξη με χαμηλή χρήση άνθρακα και οικονομία χαμηλής χρήσης άνθρακα. Και θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά ευθύς εξ αρχής. Η έκθεση τώρα στη συνέχεια της χωρίζεται σε τρία τμήματα. Καταρχάς θέλουμε να θέσουμε λίγο το προσκήνιο, εξετάζουμε το παγκόσμιο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ε, ε, περιβαλλοντικής πολιτικής, εξετάζουμε τις ε, τάσεις και κοιτάμε και τι πρέπει να περιμένουμε στις επόμενες δύο δεκαετίες, όπως σας είπα και προηγουμένως. Τα τέσσερα βασικά συμπεράσματα των εργασιών μας είναι τα εξή. Καταρχάς, πολιτικές, ε, περιβαλλοντικές και κλιματικές πολιτικές, ε, οι οποίες θα πρέπει να είναι φιλόδοξες, ε, πολύ καλά σχεδιασμένες και να εφαρμοστούν καταλήλως και εξετάζουμε και τα τρία στοιχεία γιατί θεωρώ ότι είναι απαραίτητα, διότι έτσι μόνο έχουμε ουσιαστικά ωφέλη στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Αφενός υπάρχει καλύτερο περιβάλλον και αυτό είναι άλλωστε και ο στόχος των περιβαλλοντικών πολιτικών, προφανώς, αλλά επίσης ενισχύεται η οικονομία μας και εδώ θα σας δώσω και κάποιες περαιτέρω πληροφορίες από αυτού και αυτό συνεισφέρει στην ευημερία και στην περιβαλλοντική υγεία. Αυτό το τελευταίο θέμα το κατανοούμε όλο ένα και καλύτερα, ε, διότι ε, έτσι αποφεύγουμε και κόστος ε, στα συστήματα υγείας, τα οποία πιέζονται όλο ένα και περισσότερο. Δεύτερον, όσον αφορά τις προόδους που έχουν επιτευχθεί και εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες ε, προκλήσεις και θεωρούμε ότι οι περισσότερες από αυτές τις προκλήσεις είναι στο επίπεδο των βασικών συστημάτων παραγωγής και κατανάλωσης στην κοινωνία τα ε, ε, ε, βασικά συστήματα τα οποία τονίζουμε είναι το σύστημα ενέργειας, μεταφορές και κινητικότητα, γεωργικό σύστημα και περιβαλλοντικά και ενεργειακά συστήματα. Οι προκλήσεις είναι να αλλάξουν αυτά τα συστήματα βάσει και των στόχων του 2050. Προκειμένου να γίνει αυτό θα πρέπει επίσης να ε, γνωρίζουμε ότι οι παρούσες πολιτικές ε, προσεγγίσεις ε, που είναι αυξητικές θα μας βάλουν στο σωστό δρόμο αλλά δεν θα επαρκούν. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει μια μεταβατική προοπτική η οποία θα ευθυγραμμίζεται για παράδειγμα με την απομάκρυνση του άκραντα άρθρακα από τα ενεργειακά μας συστήματα και το να περάσουμε σε ένα πιο κυκλικό σύστημα οικονομίας. Ε, δεν θεωρούμε όμως ότι η Ευρώπη θα πρέπει να φοβάται αυτό το θεματολόγιο, διότι προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες, κυρίως όσον αφορά την γενοτομία και όσον αφορά την ε, Ευρώπη ε, στην πρώτη γραμμή της επιστήμης και της καινοτομίας. Αυτό φαίνεται και στο επόμενο διάγραμμα χωρίς να επισέλθω σε λεπτομέρειες, διότι οι οθόνε αυτές είναι πολύ μικρές και δεν μπορείτε να δείτε σωστά τα διαγράμματα, αλλά ε, αν δείτε τις δύο κάτω γραμμές, εδώ έχουμε τις τάσεις από το 2000 ε, του συνολικού ευρωπαϊκού ΑΕΠ και της συνολικής απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δύο πάνω γραμμές είναι η προστιθέμενη αξία ε, της ε, οικολογικής βιομηχανίας και η απασχόληση στην οικολογική βιομηχανία. Από το 2000 έχει υπάρξει μια ανάπτυξη από το 2,8 στις 4,1 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Ε, η προστιθέμενη αξία αυξήθηκε σημαντικά, η ανταγωνιστικότητα του συγκεκριμένου κλάδου έχει αυξηθεί. Επομένως, δεν πρόκειται για ένα τομέα ο οποίος έχει επιβιώσει τις κρίσεις καλά, πρόκειται για ένα τομέα ο οποίος έχει ε, αυξηθεί παρά το γεγονός ότι υπάρχει ύφεση στην Ευρώπη. Τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης είναι ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις τρεις βασικές προτεραιότητες του εβδόμου προγράμματος για το περιβάλλον, δηλαδή να προστατεύσουμε το φυσικό μας κεφάλαιο, κάτι το οποίο συνάδει και με την πράσινη οικονομία και αυτό που αποκαλούμε πλέον λύσεις με βάση τη φύση. Αν θέλουμε να έχουμε ισχυρείς λύσεις, πρέπει να έχουμε μια ισχυρή φύση και το σχετικό κεφάλαιο. Δεύτερον, αποτελεσματικότητα προ του πόρου και μια οικονομία χαμηλής χρήσης άνθρακα και επίση ε, προστασία από περιβαλλοντικού κινδύνου για την υγεία. Υπάρχουν δύο βασικέ τάσεις οι οποίε αναδύονται. Καταρχά ότι είμαστε αρκετά καλοί σε ωφέλη αποτελεσματικότητα ε, ω προ την μείωση της ρήπενσης ε, και του πόρου μα, αλλά αυτό δεν έχει μεταφραστεί απαραίτητα σε ένα ισχυρότερο οικοσύστημα ε, και δεν έχουμε ποιότητα της ίδιας έκτασης. Ε, το σύστημα λοιπόν εξακολουθεί να υστερεί. Και επίσης δεν είμαστε τόσο αισιόδοξοι όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη εικόνα ε, σε σχέση με τις πιο πρόσφατες τάσεις και θα σας εξηγήσω γιατί αυτό το φυσικό μας κεφάλαιο. Εδώ θα δείτε, δεν θα επισέλθω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες, ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που είναι με πράσινο και εδώ πραγματικά ήμασταν ιδιαίτερα επιτυχεί στην καταπολέμηση της ρήπανσης, απομάκρυνση χημικών και ρήπανσης από τα ύδατα και τον αέρα. Έχουμε καλύτερη ποιότητα αέρα και υδάτων, εδώ ε, έχουμε όμως και το θέμα της ε, ε, βιοπικιλότητας των θαλάσσιων συστημάτων και των υδάτων συστημάτων και των οικοσυστημάτων. Εδώ βλέπουμε λοιπόν σαφώς που είμαστε καλοί και που είμαστε αποτελεσματικοί σε θέματα περιορισμού ρήπανσης, αλλά υπάρχουν περισσότερα προβλήματα με τη συστημική τους φύση. Η δεύτερη στήλη έχει περισσότερο κόκκινο και κίτρινο. Αυτή είναι η εικόνα για τα επόμενα 20 χρόνια και σε γενικές γραμμές, ε, και αυτό νομίζω ότι θα ε, διέπει τα πάντα, δύο βασικά προβλήματα δημιουργούν προβλήματα. Το ένα είναι η κλιματική αλλαγή που δυσχεραίνει όλα τα υπόλοιπα ζητήματα και ε, η απώλεια φυσικού κεφαλαίου, δηλαδή την ποιότητα των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που λαμβάνουμε από αυτά. Και οι βασικοί λόγοι για τους οποίους είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα είναι ότι οι συστημικές πιέσεις δεν μειώνονται απαραίτητος και δεύτερον είναι όλο ένα και περισσότερο παγκόσμιας φύσεως. Η δεύτερη προτεραιότητα έχει τα ίδια λίγο πολύ ε, ε, αποτελέσματα Είμαστε πολύ καλοί σε αποτελεσματικότητα. Βλέπετε ότι έχουμε περισσότερο πράσινο και κίτρινο εδώ στην πρώτη στήλη. Αλλά αν πάμε στο μέλλον, κοκκινίζουν και πάλι τα χρώματα και αυτό σχετίζεται και πάλι με την κλιματική αλλαγή και την ε, παγκόσμια υποβάθμιση του φυσικού κεφαλαίου, κάτι το οποίο πλήττει ε, και την Ευρώπη η μεγάλη επιτυχημένη ιστορία εδώ νομίζω είναι ότι χρησιμοποιούμε λιγότερη ενέργεια στην Ευρώπη πλέον. Είμαστε ε, πολύ πιο αποτελεσματικοί ως προς τη ενέργεια σε κάθε οικονομικό αποτέλεσμα. Χρησιμοποιούμε λιγότερους πόρους. Έχουμε αυξήσει την οικονομία μας από το 1990 κατά 14% μειώνοντας κατά 20% τα αεραία φαινομένα του θερμοκηπίου. Αλλά η πρόβλεψη σε παγκόσμια κλίμακα όσον αφορά τη βιοποκυλότητα, το φυσικό απο, ε, κεφάλαιο και την απώλειά τους ε, ε, λόγω της κλιματικής αλλαγής δεν είναι τόσο θετική. Όσον αφορά την προφύλαξη από περιβαλλοντικούς κινδύνους ε, για την υγεία μας, ε, στο πράσινο είμαστε στην ποιότητα των υδάτων και τις περιβαλλοντικές συνέπειες. Όσον αφορά τα αστικά συστήματα και πιέσεις, για παράδειγμα, από τις μεταφορές ε, εντός των συστημάτων αλλά και την κλιματική αλλαγή και τους νέους χημικούς κινδύνους, είμαστε στο κόκκινο και στο κίτρινο. Η πρόβλεψη εδώ και πάλι σχετίζεται κυρίως όπου έχουμε κόκκινο με την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της. Κάτι που περιμένουμε για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Σε σύνολο έχουμε εδώ αυτό το πιάνο, έχουμε αυτή την κλίμακα. Ε, αν δείτε πάνω, βλέπετε ότι υπάρχουν αρκετά πράσινα και κίτρινα πλήκτρα και θα παρατηρήσετε ότι τα περισσότερα πράσινα και κίτρινα είναι τα ωφέλη που έχουμε ως προς την αποτελεσματικότητά μας. Το κόκκινο είναι εκεί που υπάρχουν τα πιο συστημικά προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με την υποβάθμιση του φυσικού κεφαλαίου και την ε, κλιματική αλλαγή. Η πρόβλεψη για τα επόμενα 20 χρόνια δεν είναι τόσο θετικά εκεί, αλλά υπάρχουν δύο καλά στοιχεία. Πρώτον είναι ότι το μέλλον δεν πρέπει να είναι απαραίτητα συνέχεια του παρελθόντος, Επομένως, ε, ε, αυτό είναι πρόβληψη αν δεν αλλάξουμε τίποτα. Και το δεύτερο είναι ότι αυτό το παρουσιάζω στους πολιτικούς ηθήνοντες και οι πολιτικοί ηθήνοντες μπορούν να παρέμβουν. Αυτό κάνετε και επομένως μπορείτε να χρωματίσετε το, το μέλλον με πιο κίτρινο και πράσινο και όχι με κόκκινο. Ε, παρεπιπτόντως το ίδιο θα πω και θα το κάνω όταν ε, ε, μιλώ σε μεγάλους βιομηχανικούς κλάδους και στον ιδιωτικό τομέα γιατί και αυτοί χαράσουν πολιτική για το τι παράγουν και πώς το παράγουν επομένως θα μπορούσαν και αυτοί να χρωματίσουν το μέλλον με διαφορετικό τρόπο. Τώρα, ε, το γεγονός ότι αλλάζει το παγκόσμιο πλαίσιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Καταρχάς υπάρχουν πιέσεις και εκτός Ευρώπης. Αν η Ευρώπη θέλει να είναι ανταγωνιστική από πλευράς οικονομίας, δεν μπορούμε να το κάνουμε με άφθονους και φθηνούς ε, φυσικούς πόρους, γιατί δεν έχουμε σε μεγάλο βαθμό τέτοιου πόρους. Αν δείτε πόσες κρίσιμες πρώτες ύλες ε, έχουμε στον κατάλογο που έχουν ετοιμάσει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ελάχιστες από αυτές ε, βρίσκονται στην Ευρώπη, περισσότερες είναι στην Κίνα, στη Βραζιλία, στο Κονγκό, στην Τουρκία, Τουρκία και σε άλλες χώρες. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί και κυκλικοί ως προς τη χρήση των πόρων μας. Επίσης, οι πιέσεις εκτός Ευρώπης ε, είναι πολύ πιο σημαντικές και για την ποιότητα του αέρα, ε, την ποιότητα των υδάτων κλπ. Τα όρια του πλανήτη μας, που είναι το δεύτερο τμήμα ε, του τίτλου, για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για το περιβάλλον σημαίνει ότι καταλαβαίνουμε πολύ καλά τους περιορισμούς που έχουμε. Αυτό σημαίνει ότι στις διεθνές διαπραγματεύσεις προκειμένου να πείσουμε ε, τους εταίρους μας να συμμετέχουν για να μετριάσουμε τις συνέπειες για το κλίμα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και επομένως θα πρέπει να υπάρχει ένα καλό ε, καθορισμένο πλαίσιο και μια πολύ φιλόδοξη ευρωπαϊκή πολιτική ως σημείο κίνησης. Βεβαίως υπάρχουν πολλά περίπλοκα στοιχεία, μεγάλη αβεβαιότητα και ε, αλληλεξαρτήσεις μεταξύ περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών ε, πτυχών. Τώρα, για να μην καθυστερήσουμε, θα παραλείψω κάποιες διαφάνειες και θα περάσω σε αυτήν. Κάποιοι από εσάς μπορεί να την έχετε δει. Όταν ε, αναφερόμαστε στο μέλλον της πολιτικής ε, και το τι διαφορά υπάρχει μεταξύ των επικεντρωθούμε σε αυξητικά ωφέλη των ε, όσων έχουμε αυτή τη στιγμή και να μην επικεντρωθούμε στην καινοτομία, ε, νομίζω ότι αυτή η εικόνα μας δείχνει πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί στις μηχανές καύσης ε, και η ευρωπαϊκή βιομηχανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στο τομέα αυτό. Αν θέλουμε όμως το σύστημα μεταφορών και κινητικότητας να είναι χωρίς άνθρακα, σημαίνει ότι χρειαζόμαστε διαφορετικά στοιχεία και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ένα από τα στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξουμε τεχνολογία, κυρίως διότι οι κοινοτήρε αυτών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα είναι με διαφορετική χρήση ενέργειας. Εάν όμως όλοι οδηγούμε αυτό το ίδιο αυτοκίνητο με τον ίδιο τρόπο που κάνουμε και τώρα, με τον ίδιο χρόνο, κατά πάσα πιθανότητα ο καθένας μόνος του. Και ταυτόχρονα κατεβαίνουμε από την οδό Λουά, από τη Σουμάν και είμαστε όλοι κολλημένοι στην κίνηση, δεν θα αλλάξει η κυκλοφοριακή συμφέρηση και επίσης ε, θα χρησιμοποιούμε άλλους πόρους, γιατί και οι μπαταρίες χρειάζονται χρήση πόρων. Η αλλαγή λοιπόν που σκεφτόμαστε σε συστημικό επίπεδο είναι να σκεφτούμε τι απαιτήσει θα υπάρχουν για την κινητικότητα, να σκεφτούμε λίγο και θέματα χωροταξίας ε, και το συνδυασμό του εργασιακού ε, και του προσωπικού βίου, τι θα κάνουν τα παιδιά μας ε, και έτσι θα κατανοήσουμε λίγο καλύτερα το σύστημα κινητικότητας. Σαφώς και το αυτοκίνητο θα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και σίγουρα χρειαζόμαστε ένα αυτοκίνητο που θα έχει μηδενικές εκπομπές, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το σύστημα και να κατανοήσουμε το σύστημα και όχι να αντικαταστήσουμε τον κινητήρα στο ίδιο σύστημα. Τώρα, ο πρόεδρος μου δείχνει το ρολόι του, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τελειώνω. Για το μέλλον λοιπόν, όταν επενδύουμε σήμερα σε αυτά τα μακροπρόθεσμα ωφέλη και στόχους, ε, αντιλαμβανόμαστε ότι οι ανάγκες που έχουμε σε επενδύσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αλλά οι επιλογές που θα κάνουμε σήμερα θα έχουν και συνέπειες μακροπρόθεσμα. Όταν επενδύουμε σε ένα σύστημα ε, κινητικότητας και μεταφορών σήμερα, θα είναι το ίδιο σύστημα το οποίο θα λειτουργεί ακόμα και το 2050. Ανάλογα λοιπόν με τις επιλογές που θα γίνουν σήμερα, θα καθορίσουμε με ποιο τρόπο θα φτάσουμε στους στόχους του 2050 ή δεν θα τους επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Επίσης πρέπει να αντιληφθούμε ότι ήδη επενδύονται τεράστια ποσά και πόροι ε, στην οικονομία του σήμερα. Επομένως, η σωστή κατεύθυνση αυτών των πόρων είτε θα προέρθουν από το ορίζοντα 2020, είτε θα προέρχουν από το ε, Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, είναι πολύ σημαντική. Και βάσει της έκθεσή μας θεωρούμε ότι αυτές οι επενδύσεις σε μια πράσινη οικονομία θα πρέπει να πηγαίνουν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και αυτό σημαίνει χωρίς άνθρακα, κυκλική οικονομία και σχετικές θέσεις εργασίας οι οποίες συνοδεύουν αυτή την οικονομία. Και αυτές είναι οι κατάλληλες επιλογές. Τα συστήματα, ε, ε, το οικοσύστημα μάλλον και τα όρια του πλανήτη μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αν θέλουμε να έχουμε μια οικονομία που βασίζεται στη βιολογία και στη φύση δεν μπορούμε να έχουμε έχουμε ε, αλλαγές οι οποίες ε, δεν θα μας επιτρέπουν να έχουμε καλή υγεία και ευημερία. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τις πιέσεις στα ασφαλιστικά συστήματα και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τώρα, η αλλαγή της φορολόγησης και ε, η σταδιακή απουσία χρήσης επιδοτήσεων που είναι ζημιογόνες για το περιβάλλον μπορεί να δώσουν κίνητρα για επενδύσεις και καινοτομίες. Ε, ελάχιστες χώρες όπως η Πορτογαλία για παράδειγμα έχουν επενδύσει σε ε, τέτοια πράγματα και οι επιδοτήσεις για τα περιβαλλοντικά ζητήματα παρακολουθούνται όλο ένα και περισσότερο και εμείς ε, στον οργανισμό μας τα παρακολουθούμε τα θέματα αυτά. Εδώ είναι η τελευταία διαφάνεια. θεωρούμε ότι προκειμένου να επιτευχθεί το όρεμα του 2050 βάσει των όσων κατανοούμε και των τάσεων που υπάρχουν είναι δυνατό, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση όσον αφορά τις δράσεις και τις επενδύσεις που πρέπει να κάνουμε σήμερα. Και γι' αυτό και ακριβώς θεωρούμε ότι ε, επενδύσεις ε, όπως το Στρατηγικό Ταμείο Επενδύσεων και κάποιες άλλες επενδύσεις ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κυρίως αν θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένη κατεύθυνση για να επιτύχουμε το όρομα του 2050. Όσον αφορά τις συστημικές αλλαγές θεωρούμε ότι εδώ θα πρέπει να υπάρχουν ευκαιρίες για αξιοπρεπή εργασία και δικαιοσύνη και να γίνουν σεβαστά και τα περιβαλλοντικά όρια διότι το περιβαλλοντικό θεματολόγιο δεν είναι ένα θεματολόγιο αυτούσιο, αν είναι ένα θεματολόγιο παραγωγής και κατανάλωσης, βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινωνίας και όχι στο περιθώριο. Ε, και θα πρέπει να υπάρχει αξιοπρεπής απασχόληση, διότι και αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο. Ε, ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρχουν αποτελέσματα. Επίσης, θεωρούμε ότι η έκθεσή μας καταδεικνύει ότι η Ευρώπη ε, εδώ και τέσσερις δεκαετίες οικοδομεί την ισχυρότερη περιβαλλοντική πολιτική στον πλανήτη έχει ε, αποφέρει καρπούς για τους Ευρωπαίους πολίτες αρκετά καλά, με αρκετούς τρόπους, αλλά αν μπούμε σε ένα νέο στάδιο ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, το οποίο επικεντρώνεται περισσότερο σε αυτούς τους κρίσιμους στόχους ε, μιας κυκλικής οικονομίας χαμηλής χρήσης άνθρακα και ε, καλύτερης προσαρμοστικότητας και αντοχής, θα δημιουργήσουμε πολύ καλύτερες ευκαιρίες για την Ευρώπη. Δεν πρόκειται για απειλή, πρόκειται για ευκαιρία. Διότι το λογικό ερώτημα, και εδώ θα σταματήσω κύριε Πρόεδρε. Όταν δίνουμε ε, ερωτήματα που αφορούν με τη λογική, ε, είναι λογικό για παράδειγμα από το 80 να πάμε στο 95% μείωση των εκπομπών αέριου του θερμοκηπίου. Είναι λογικό να ζητούμε από τις επιχειρήσεις να σκέφτονται κυκλικά και όχι γραμμικά. Εμείς θεωρούμε ότι είναι οι μόνες λογικές επιλογές, διότι εάν δεν αλλάξουμε κατεύθυνση, ε, υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να καταλήξουμε εκεί που επιθυμούμε. Και ξέρουμε ότι τα παρόντα συστήματα παραγωγής και κατανόλησης δεν είναι βιώσιμα μακροπρόθεσμα και επομένω αν συνεχίσουμε προς αυτό το δρόμο είναι παράλογο. Το λογικό είναι να κατευθυνθούμε προς μια διαφορετική ε, κατεύθυνση και νομίζω ότι η έκθεση αποδεικνύει πολύ καλά γιατί ε, η κατεύθυνση του πακέτου για το κλίμα και την ενέργεια της κυκλικής οικονομίας και του 7ου προγράμματος για το περιβάλλον είναι η καλή λύση για να ξεφύγουμε από την κρίση όχι μόνο ισχυρότερη αλλά προετοιμασμένη και για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα ε, και όχι τις προκλήσεις του παρελθόντος. Σας ευχαριστώ. Ξεκινάμε αμέσως τη συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Φαρία, που είναι ο αξιωματούχο ε, επαφής με την υπηρεσία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να καλωσορίσω τον κύριο Μπρένινγκ, τον Διευθυντή, τον κύριο Σκούλος και τον κύριο Χέι. Επίσης να συγχαρώ την ε, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, ιδιαίτερα τον Διευθυντή, για το εξαίρετο έργο που μας παρουσίασε. Η έκθεση που μας υποβάλλεται σήμερα δείχνει την πρόοδο που έχουμε υλοποιήσει σε σχέση με το περιβάλλον στην Ευρώπη. Βέβαια έχουμε στόχους που δεν έχουμε ακόμη υλοποιήσει και αυτό και χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέσυρε σημαντικά πακέτα, όπως είναι το θέμα των αποβλήτων και της ε, ποιότητας του αέρα. Ε, απέσυρε αυτά τα πακέτα για να τα αναδιατυπώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί, για ποιους ακριβώς λόγους ε, το έκανε. Για μερικές πτυχές θα γίνουν μεταρρυθμίσεις. Ελπίζω οι μεταρρυθμίσεις αυτές να καταστήσουν προτάσεις πιο φιλόδοξες και πιο αποτελεσματικές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο Ιβο Μπέλετ τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση αλλά θα την υποβάλω στα Ολλανδικά κύριε Μπρέινιγκς. Ε, βεβαίως μας απασχολεί το κλίμα και το σύστημα εμπορίας εκπομπών όπως είπατε και ξέρετε κύριε Μπράνιγκς και βεβαίως πρέπει να το ε, επισκευάσουμε αν θέλετε με το απόθεμα σταθερότητας. Βεβαίως όταν μιλάμε για βιομηχανία θα πρέπει να δούμε το τι θα γίνει με τις ε, πιθανές εξελίξεις ε, στο μέτωπο της διαρροής του άνθρακα. Ποιο μήνυμα έχετε εσείς λοιπόν για τις επιχειρήσεις ε, έντασης ενέργειας που αντιμετωπίζουν πάρα πολύ έντονο ανταγωνισμό, ειδικά όσον αφορά το έμεσο κόστος, το κόστος της ενέργειας και του διοξιδίου του άνθρακα που πρέπει να πληρώσουν δεδομένου του ότι το κόστος της ενέργειας στη ΣΥΠΑ είναι κλάσμα αυτού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να μας ε, πείτε κάτι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκρότα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. συζητάμε πάρα πολύ για αυτά τα θέματα και με τον κύριο Κατάινεν ε, για το πώς θα δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας. Τα νούμερα είναι σαφή δημιουργούνται θέσεις εργασίας ε, στις νέες τεχνολογίες, ε, τις ανανεώσιμες ενέργειες. Οπότε θεωρώ πως θα πρέπει να δώσουμε βάρος ε, και στο ζήτημα της κυκλικής οικονομίας. Μιλάμε, μιλάμε εδώ πέρα πάρα πολύ για την TTIP στο Κοινοβούλιο, την Διαταδική Εμπορική Συμφωνία και το τι δυνατότητες μας δίνει. Πήγαμε και με μια αντιπροσωπεία στη ΣΥΠΑ για το θέμα αυτό και συναντήσαμε τους ομολόγους μας που ήταν κάπως συγκρατημένοι Τώρα εμείς την TTIP την βλέπουμε 2017-18 και αν. Λοιπόν, αν ε, συγκρίνουμε αυτά τα δύο, δηλαδή δυνατότητες για θέση εργασίας με μια κυκλική οικονομία, τι μας λέει η, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, πού οδηγεί αυτός ο δρόμος. Το ερώτημα του Ιβομπέλετ ήταν πάρα πολύ καλό, η διαρροή άνθρακα, η λεγόμενη, ε, που συχνά την ακούμε αλλά συχνά μπερδευόμαστε κιόλας γιατί έτσι δεν περιλαμβάνεται και το έμεσο κόστος των επιχειρήσεων. Τι συμβουλή μπορείτε να μας δώσετε λοιπόν για να λάβουμε υπόψη στους κανόνες περί ανταγωνισμού αυτό το έμεσο κόστος και το πρόβλημα αυτό. Όσον αφορά τώρα την ηλεκτρική κινητικότητα καλά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά αν ο ηλεκτρισμός ε, παράγεται από άνθρακα, ε, καλύτερα να καίνε βενζίνη, γιατί τελικά εκπέμπουν λιγότερους ρήπους ε, από ότι ο ηλεκτρισμός που παράγεται από άνθρακα. Δηλαδή μη μετατοπιστούν οι εκπομπές από την εξάτμιση του αυτοκινήτου στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας ε, πρέπει και η ηλεκτρική ενέργεια να είναι καθαρή και βεβαίως είναι κάτω στο κατασκευή. και αυτό βεβαίως συνδέεται με το θέμα της δικτύωσης και συχνά το παραμελούμε. Έξυπνα κυκλοφορία, όχι μόνο έξυπνα δίκτυα, να ε, αποφεύγουμε και τα μποτιλιαρίσματα ξέρω, τα είπα, είπα πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να τα πούμε εδώ πέρα στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ, ο κύριος Μέκερ. Ευχαριστώ. Κύριε Μπράινινγκς, σας καλωσορίζω και εξ ονόματος του ECR. Θα μιλήσω τη γλώσσα μου ε, για να συνεννοηθούμε κιόλας. Η Eurostat δημοσίευσε τα νούμερα για τα απόβλητα και την κατεργασία του το 2013 και υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και δεν μπορούμε να μιλάμε για ίσους όρους ανταγωνισμού. Ποιο είναι το όραμά σας λοιπόν για βελτίωση της εφαρμογής της σχετικής ε, νομοθεσίας και για μια ιεραρχία των ε, απορριμμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να καταλήξει στο τέλος του έτους ε, σε μια πιο φιλόδοξη πρόταση για τις ε, συσκευασίες. Θα πρέπει όμως ε, να πούμε πως στέλνουν ανάμικτα μηνύματα από πλευράς κομισιών Επίσης σωστά αναφέρατε την επίκαιρη περίπτωση των πρώτων υλών και την επισφάλεια που υπάρχει από πλευράς προμήθειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δικό σας το μήνυμα στις ε, Ευρωπαίες, ευρωπαϊκές μας επιχειρήσεις για την κυκλική αυτή οικονομία. Ευχαριστώ κύριο Γκέρμπραντι. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον κύριο Μπρένιγκς για την ε, πολύ ξεκάθαρη παρουσίαση της κατάστασης του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2015. Και σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον ε, είναι ανακούφιση για μας να βλέπουμε κάποιον που στηρίζεται σε πραγματικά περιστατικά. Και αυτή, αυτό είναι και το πλεονέκτημα της έκθεσης. Δεν περιλαμβάνει ένα πολιτικό όραμα για το μέλλον, αλλά είναι μια συμπίληση στοιχείων και πραγματικών περιστατικών. Και με βάση αυτά τα στοιχεία περιγράφει την μελλοντική μας πορεία. Το συμπέρασμά σας είναι κάπως ζωφερό θα έλεγα, κάπως απεσιόδοξο. Λέτε ότι η ανάλυση υποδεικνύει ότι ούτε από μόνες τους οι περιβαλλοντικές πολιτικές, ούτε ε, τα κέρδη της αποτελεσματικότητας από την οικονομία θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε το στόχο μας για το 2050. Με άλλα λόγια, ό,τι και αν κάνουμε σήμερα, πόρο απέχουμε από την υλοποίηση των μελλοντικών μας στόχων. Και αν αυτό το συνδέσω με το γεγονός ότι οι κατευθυντήριε γραμμές πολιτικής του Προέδρου Γιούνκερ δεν αναφέρουν πουθενά κανένα από αυτά τα στοιχεία της έκθεσης, δεν κάνουν οποιαδήποτε τέτοια μνήμα, διαπιστώνω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτικών και των πραγματικών στοιχείων που στοιχειοθετούν την έκθεσή σας. Οπότε η, έκθεση, η, η ερώτησή μου απευθύνεται περισσότερο στον πρόεδρο παρά στον κύριο Μπρόνιξ. Μήπως θα έπρεπε η συζήτηση που θα οργανώσουμε στο μέλλον θα πρέπει να τη χάνει τη παρουσία του, του Πρόεδρου Γιούνκερ και όχι του Επιτρόπου Βέλα. Γιατί χρειάζονται ρηξικέλευτε μεταρρυθμίσει και καλό θα ήταν να γίνει σε μια κανονική συζήτηση τη Ολομέλη Επιτροπή παρουσία του Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και για την ερώτηση. Ο κύριο Μαζή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και να επενέσω ε, το εμπεριστατωμένο πόνημά του. Μερικές φορές η διάβια μας κάνει απεσιόδοξους, αλλά η βούληση δράσης μας υποχρεώνει σε μια αισιοδοξία. Γι' αυτό και θα υποβάλω μια ερώτηση, γιατί φοβάμαι ότι το σύνολο των δημοσίων πολιτικών που εφαρμόζουμε φοβάμαι ότι θα, θα αποτύχει, θα προσκρούσει σε πολιτιστικά προβλήματα. Διερωτώ με λοιπόν, οι ε, ανθρωπιστικές επιστήμες ε, συνεκτιμώνται, συνεκτιμώνται στην ε, όλη αυτή τη συζήτηση για το περιβάλλον. Γιατί νομίζω ότι η έννοια της ευτυχίας, η σχέση που έχουμε με το χρόνο ή η σημασία που αποδίδουμε στο άτομό μας, όλα αυτά τα θέματα επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο δεχόμαστε τις διάφορες πολιτικές. Δεύτερον, η ημερομηνία που μας αναφέρατε είναι το 2050. Το 2050 θα έχουμε 9 δισεκατομμύρια κατοίκους στον πλανήτη μας. Και εμείς ε, θα χάσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 90 εκατομμύρια κατοίκους με βάση τους υπολογισμούς στο ΙΕ. Οπότε οι λύσεις ε, ε μερικές φορές βρίσκονται και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις δράσεις μας για να είναι κοινέ. Επίση, ό,τι αφορά τη γαλάζια οικονομία, θεωρώ ότι ο ρόλος τη γαλάζιας οικονομία μπορεί να είναι σημαντικός, υπό τον όρο ότι θα θέσουμε από τώρα κάποια μέτρα, γιατί δυστυχώς ε, έχουμε, ε, έχουμε καταφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στις διάφορες ε, στους, σε διάφορες ε, γεές και εδάφη. Ελπίζω να μην έχουμε τις ίδιες ανεπανόρθωτες βλάβες και στον πυθμένα των ε, ωκεανών. Η κυρία Τσεγκερέκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεδρίαση και συνάντηση χτες, αλλά κάποια πράγματα δεν ε, ξεκαθάρισαν. Χτες μας είπε ο επίτροπο Ποσυνατούρα η Natura θα έχει 200 εκατομμύρια ευρώ. Έχω μια ερώτηση όμως. Πώς θα γίνει αυτό, γιατί πραγματικά είμαστε στην πρωτοπορία στην Ολλανδία, στις περιοχές Natura, αλλά το γεγονός είναι πως δεν λαμβάνεται υπόψη ο άνθρωπος. Θα πρέπει πράγματι τα χίλια είδη ε, ζώων και φυτών να αναπτυχθούν και έχουν και μια ζώνη προστασίας αρκετών ε, χιλιόμετρων αλλά οι αγρότες δεν ε, έχουν ε, καμία βοήθεια, χρειάζονται να υποβάλουν ειδικέ αιτήσει για να λάβουν άδεια για περιβαλλοντικές δραστηριότητες οι οποίες κοστίζουν πάρα πολύ το συγκεκριμένο ερώτημα. Μήπως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις ε, κοινωνικο-περιβαλλοντικές ε, ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Ναι, οπωσδήποτε την φύση, αλλά κάπου πρέπει να υπολογίσουμε και τον άνθρωπο. Υπάρχουν αγρότες οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα 800 χρόνια, καλλιεργούν τα ίδια φυτά 800 χρόνια και ε, δεν τους επιτρέπεται να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο ε, φυτό. Εντάξει, συμφωνώ, περιβαλλοντική πολιτική, αλλά κάπου πρέπει να έχει και μια ευκαιρία και ο άνθρωπος να ζήσει. Σας ευχαριστώ, κυρία Γκουτλάντ. Ε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω την μητρική μου γλώσσα. Ευχαριστώ τον κύριο Μπράινινγκς για την πάρα πολύ καλή παρουσίαση που έκανε. Πρέπει να πω πως ε, πραγματικά είχε πάρα πολλές ε, πληροφορίες. Και οπωσδήποτε θα στείλουμε και τις σχετικές ε, ερωτήσεις στην γραμματεία αν δεν απαντηθούν. Αλλά πρώτα απ' όλα κάποιες ερωτήσεις σε εσάς. Έχουμε τους διάφορους ε, κλάδους που αναφέρατε και την ανάπτυξή τους. Ε, ε, μιλήστε για μια αύξηση 208%. Υπάρχουν συγκεκριμένοι όμως κλάδοι εντός της οικονομίας αυτής που αναπτύχθηκαν πιο δυναμικά. Μετά, μιλήσατε για το περιβάλλον ε, στην ε, πολεοδομία, στην χωροταξία μάλλον ε, καλύτερα και είπατε πως αν είναι να γίνει κάτι για το 2050 πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα. Έχετε κάποια συγκεκριμένα πράγματα στα οποία θα θέλατε να ασκηθεί περισσότερη πίεση μετά. Κάθε πέντε χρόνια υποβάλλεται αυτή η έκθεση. Υπάρχουν κάποιοι τομείς, κάποια ευρήματα τα οποία σας προξένεξαν εντύπωση και στα οποία πρέπει να αντιδράσουμε ιδιαίτερα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κάτι το οποίο με απασχολεί. Οι μέλισσες ε, που διαπιστώνουμε σε διάφορες χώρες ότι πεθαίνουν και έχουμε βεβαίως την επίδραση ενός κοκτέιλ φαρμάκων ε, ζυζανιοκτώνων κατά βάση παρά το ότι υπάρχει ένα μορατόριουμ για τη χρήση των ουσιών αλλά πολλές από αυτές ε, τις ουσίες επηρεάζουν τις μέλισσες οι οποίες μετά πεθαίνουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε κάτι γιατί οι μέλισσες είναι σημαντικές για τον άνθρωπο και πρέπει και αυτές να επιζήσουν. Επίσης, και η αρχή βεβαίω ε, των χημικών πρέπει να κάνει κάτι. Ευχαριστώ κύριο Σλέκ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, πολύ αξιόλογη αυτή έκθεση και θα πρέπει να τη στείλετε σε όλους τους πρωθυπουργού ε, των κρατών μελών για να λάβουν από πρώτο χέρι πληροφορίες για το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και πώς μπορούμε από κοινού να υλοποιήσουμε τους στόχους της περιβαλλοντικής αυτής πολιτικής. Έχω τρεις ερωτήσεις. Έχουμε δύο διαφορετικά προβλήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το πρώτο είναι πώς θα πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτεί πολύ σοβαρά στο μέλλον το θέμα της κυκλικής οικονομίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, γιατί θα δημιουργήσουν και οικονομική ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης, όπως επισημαίνεται και στην έκθεσή σας. Και το δεύτερο είναι πώς θα ε, εμπλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας σε αυτή τη διαδικασία. Στις ιστοσελίδες ε, του οργανισμού περιβάλλοντος ε, βρήκα δύο πολύ σημαντικές ε, εφαρμογές. Το ένα αφορούσε τη μόλυνση ε, του περιβάλλοντος και τέτοιου είδους εφαρμογές θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πιο εντατικά για να μπορούμε να στέλνουμε αυτές τις πληροφορίες στο ευρύ κοινό. Επίσης υπάρχει μια άλλη εφαρμογή που δίνει πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα. Αλλά δυστυχώς δεν έχετε πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα για όλες τις χώρες μέλη. Γιατί, γιατί λείπουν αυτές οι πληροφορίες για ορισμένες χώρες. Δεν έχουν ε, monitoring οι χώρες αυτές, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν αυτές τις πληροφορίες ή δεν σας τις στέλνουν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Πολύ σημαντικές αυτές οι δύο εφαρμογές που έχετε σκοπεύετε να περιλάβετε και άλλες ε, εφαρμογές στις ιστοσελίδες σας, γιατί ιδιαίτερα οι νέοι χρησιμοποιούν πολύ τα κινητά και τις νέες τεχνολογίες. Καλό θα ήταν λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να διαδώσουμε αυτές τις γνώσεις και να αφυπνίσουμε τους ε, συμπολίτες μας και τους νέους που ενδιαφέρονται περισσότερο για αυτές τις τεχνολογίες για τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Ευχαριστώ τον ε, Διευθυντή του Οργανισμού Περιβάλλοντος για την εξαιρετική ε, ε, παρουσίαση. Το 2015 είναι το διεθνές έτος του εδάφους. Δόθηκε σημασία σε ένα πόρο ο οποίος δεν είναι ανανεώσιμος και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος στην έκθεση για το περιβάλλον στην Ευρώπη λέει ότι τα ε, επίπεδα διαβροφοποίησης του εδάφους, ε, υποβάθμιση και μόλυνσης των οργανικών υλών δείχνουν όλα ότι μειώνονται οι δυνατότητες που έχει το έδαφος. Η έκθεση λέει ότι μια συνεκτική ευρωπαϊκή πολιτική για το έδαφος θα μας δώσει τη δυνατότητα να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας και να εποπτεύουμε με αποτελεσματικό τρόπο την κατάσταση του εδάφους και να καταπολεμήσουμε και τη ρήπανση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν έχει μια στρατηγική για τα εδάφη παρά το γεγονός ότι η προστασία του είναι πάρα πολύ σημαντική για να έχουμε ένα υγιές περιβάλλον στην Ευρώπη. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 2006 μπλοκαρίστηκε από μια μειοψηφία κρατών μελών. Αλλά επειδή είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, δεν θεωρείτε εσεί ότι θα πρέπει να ξαναπροταθεί μια στρατηγική για τα εδάφη και σε περίπτωση που μπλοκάρουν και πάλι μια μειονότητα κρατών μελών θα μπορούσε να εγκριθεί μέσω ενισχυμένη συνεργασία. Να τονίσω επίσης και το εξή. Εγώ συμφωνώ όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων, συμφωνώ ε, με τα όσα ακούστηκαν προηγουμένως από τον συνάδελφο Ματίας Γκρότε. Εάν θέλουμε να αντικαταστήσουμε την παραδοσιακή μορφή κίνησης με ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μετά χρησιμοποιούμε άνθρακα για να κινηθούν αυτά τα αυτοκίνητα, είμαστε σε δυνότερη θέση από ό,τι πριν. Και επίσης θα ήθελα να προσθέσω και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Αν αυτή την ενέργεια τώρα την ε, ε, συγκεντρώνουμε με τις παρούσες μπαταρίες, για τις οποίες προβλέπονται και απαιτούνται εξόριξη ε, ε, υλών που είναι ακόμα πιο καταστροφικές για το περιβάλλον, σίγουρα καταστρέφουμε ακόμα περισσότερο το περιβάλλον από ό,τι στο παρελθόν. Πρέπει να αντικαταστήσουμε με βιώσιμα μοντέλα, τα οποία πραγματικά θα είναι γαλάζια, όχι μόνο γιατί έχουν ως ε, σημείο αναφορά στη θάλασσα, αλλά και τη βιωσιμότητα, τα φυσικά οικοσυστήματα. Αυτά είναι αυτά τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε μια πραγματική μετάβαση προς το μέλλον. Ευχαριστώ κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, το έγγραφο αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και θα είναι πολύ χρήσιμο για μας ε, όλους. αν κατάλαβα καλά, το σχέδιο για το 2050 είναι ευημερία για τον πλανήτη μας ε, με το 7ο πρόγραμμα ε, δράσης για το περιβάλλον, αλλά φυσικά όλα αυτά δεν θα πρέπει να μείνουν κενό γράμμα. Ε, καταλαβαίνουμε ότι όλοι ανθίστανται στις αλλαγές, καταλαβαίνουμε τι δυσκολίες μπορεί να υπάρχουν βραχυπρόθεσμα ε, και για το οικονομικό και βιομηχανικό περιβάλλον, διότι τα πάντα μεταφράζονται σε οικονομία προφανώς. Εγώ θα ήθελα να θίξω το θέμα της χρηματοδότησης. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα, σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση. η ε, δεν θα λειτουργήσει. Επομένως, ε, ε, χρηματοδότηση από το δημόσιο όταν πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν πια χρήματα και δεν μπορούν να επενδύσουν, ε, πραγματικά μας δημιουργεί δυσκολίες. Πώς μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα και την ποιότητα των υδάτων. Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα ε, Εμένα δεν με ανησυχεί η ρήπανση από τα αυτοκίνητα. Πιστεύω ότι στην επόμενη δεκαετία θα έχει προχωρήσει η τεχνολογία, θα έχουμε νέε και πράσινε τεχνολογίε. Η ρήπανση από τα αυτοκίνητα δεν με ανησυχεί λοιπόν. Η ρήπανση όμω από τι βιομηχανίε, από το αστικό περιβάλλον, η επιστροφή στην ενέργεια του άνθρακα. Αυτά είναι καταστροφή και φυσικά δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτή την ενέργεια. Σίγουρα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα, αλλά και ε, για ε, καθαρές τεχνολογίες και ε, εδώ χρειαζόμαστε επενδύσεις. Πώς θεωρείτε λοιπόν ότι μπορούμε να επηρεάσουμε και τα κράτη-μέλη μέσω φορολόγησης, πράσινης φορολόγησης, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, ώστε να λάβει υπόψη όλες αυτές τις επενδύσεις Αναφερθήκατε επίσης και στο Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Συμφωνώ. Εσείς πώς βλέπετε όμως ε, το θέμα, τι προσανατολισμό πρέπει να έχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μπάλας. Θα είμαι σύντομος. Ε, θα ήθελα να σταθώ σε ένα στοιχείο την ένταση που υπάρχει μεταξύ ε, της εκβιομηχάνησης της Ευρώπης και τον οικολογικό τομέα. Υπάρχει ένας τομέας που θα μπορούσε να συμφιλειώσει τα δύο. Στην ενέργεια είναι περίπλοκα παρά το γεγονός ότι εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Είναι ο τομέας της κυκλικής οικονομίας. Γιατί η κυκλική οικονομία σήμερα είναι ένα από τα μέσα που μας επιτρέπει να πούμε ότι ένα ε, προϊόν θα έχει ε, περισσότερες οικονομικές ζωές και κάθε φορά θα υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης, ε, παραγωγής, επομένως χώρος εργασίας, ε, παραγωγής και εργασίας, τεχνολογίες που θα είναι χρήσιμες για όλους, που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και θα δώσουν νέα δυναμική σε κάποιες περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι ένα και λιγότερο ανταγωνιστικές λόγω της παγκοσμιοποίησης. Από αυτή την άποψη υπάρχει μια οδηγία η οποία ε, σήμερα χάθηκε. Ο κύριος Τίμερμανς δεσμεύτηκε να κάνει κάποιες προτάσεις στο τέλος του έτους επί του ζητήματος. Η οδηγία αυτή <coughs> αφορούσε το θέμα της ανακύκλωσης των απορριμμάτων αλλά και την οικολογική αντίληψη, το eco-conception. Ε, μπορείτε να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα για το θέμα αυτό. Ξέρω ότι δεν είστε αυτός που λαμβάνει τις αποφάσεις, αλλά θα μπορούσατε να μας ευκρινίσετε κάποια πράγματα. Και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο ε, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό και να απαιτήσει να υπάρχουν ε, ε, ταχύτατα δεσμεύσεις, διότι αν πρέπει να υπάρχει κάποια σχέση ε, σε θέματα πράσινης βιομηχανίας, είναι σε αυτά τα θέματα και δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι αυτά είναι αντιφατικά. Ευχαριστώ κύριε Γκζιμπ. Ευχαριστώ κύριε Πράδρα. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που παρουσίασε και που δημοσίευσε, είναι δημοσιευμένη και μπορεί ο καθένας να τη διαβάσει. Και πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε, κύριε Διθεντά, ότι κρίσιμα κοιτάσματα ε, σημαντικών πρωτονυλών βρίσκονται εκτός Ευρώπης. Οπότε θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη στη στρατηγική μας για τις πρώτες ύλες. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία είχαμε μία έκθεση για τις σπάνιες γέες. Και μάλιστα το 80% σχεδόν αυτών των σπανίων γεών βρίσκονται στα χέρια μιας χώρας. Κάτι άλλο σημαντικό είναι το ζωηρό ενδιαφέρον για αποθέματα που βρίσκονται σε σημαντική σε περιοχές με, σημαντικό, ε, με σημαντική αξία οικολογική. Και δεν ξέρω πώς η, τι επιρροή θα έχουν εδώ οι επίδοξοι επενδυτές. Για παράδειγμα, τι γίνεται με τους φυσικούς πόρους της Αρκτικής. Εκεί υπάρχει σημαντικός φυσικός πλούτος και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό των ενεργειακών πόρων της Αρκτικής. Και εκεί ενδιαφέρονται χώρες που είναι εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και που πραγματοποίησαν σημαντικά βήματα σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση αυτών των πόρων. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διάρκεια ζωής των προϊόντων. Αφενός μας ενδιαφέρει αυτή η ιδέα που βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, αλλά πολύ αργά, το θέμα της κυκλικής οικονομίας. Αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι η διάρκεια ζωής πολλών προϊόντων ε, μειώθηκε. Και μερικές φορές η αλλαγή ενός πολύ μικρού ανταλλακτικού, ακόμη και σε οικιακές συσκευέ ε, είναι ασύμφορη. Μερικές φορές είναι, συμφέρει περισσότερο να αγοράσουμε ένα νέο προϊόν, να αλλάξουμε το προϊόν, παρά να αλλάξουμε ένα συγκεκριμένο ανταλλακτικό. Παρόλο που θα μπορούσε με την αλλαγή αυτή να λειτουργήσει ε, για, για, διάφορο, για καιρό ακόμη το προϊόν. Και μάλιστα η μάρκα Electrolux ακριβώς ε, ε, έχει συνδεθεί στο μυαλό μας με το σύνθημα της άριστης ποιότητας. Αλλά μερικές φορές και μικρά ανταλλακτικά είναι δύσκολο και δαπανηρό να αλλάξουν, ενώ ταυτόχρονα έχουμε πολύ μικρό απόθεμα φυσικών πόρων. Οπότε αυτό το θέμα θα πρέπει να το συνδυάσουμε, διάρκεια ζωής των προϊόντων με το θέμα της κυκλικής οικονομίας, για να χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο και να παρατείνουμε τη διάρκεια της ζωής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία TTIP, το θέμα της, του μοντέλου της κατανάλωσης αλλά και του μοντέλου παραγωγής ε, είναι σημαντικά και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και στη συμφωνία τη Διατλαντική με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, ε, ε, είναι πολύ σημαντική μια ιδέα που προτείνεται στην έκθεσή σας, προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και πέραν των μεγάλων αστικών κέντρων ώστε να περιοριστεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Δεν ξέρω αν βλέπετε κάποιους κινδύνους ή απειλές για αυτό το θέμα. Βλέπω ότι είναι έτοιμος να σηκώσει το σφυράκι του κύριος Πρόεδρος, γι' αυτό και βάζω τελεία. Okay. Σας ευχαριστώ. Πληθώρα ερωτήσεων και πολλοί συνάδελφοι υπέβαλαν ε, τις ερωτήσεις τους στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουμε δύο εκπροσώπους, τον καθηγητή Μάικλ Σκούλα και τον καθηγητή Χέι. Δεν ξέρω ποιος θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω θερμά για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε και για την ανανέωση της εντολής μας προκειμένου να εκπροσωπούμε εσάς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά για την παρουσία μου εδώ μετά από την πολύ ενδιαφέρουσα και καρποφόρα συζήτηση που έγινε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο-τρία θέματα που αφορούν το ρόλο μας στην, στον οργανισμό και την έκθεση. Πιστεύω κύριε Πρόεδρε ότι η συγκεκριμένη έκθεση για το 2015 αντικατοπτρίζει και μάλιστα με τον πιο εύστοχο και επιτυχημένο τρόπο τις προσδοκίες ε, και το πνεύμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την προσέγγιση που υιοθετεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και την ε, σωρία προβλημάτων που υπάρχουν. Και μάλιστα αυτό γίνεται με πιο συστηματικό τρόπο, με βάση πραγματικά περιστατικά, συγκεκριμένα στοιχεία και αντιμετωπίζοντας βασικά αίτια, τα θέματα παραγωγής, κατανάλωσης και τα μοτίβα παραγωγής, κατανάλωσης και ε, χρήσης των πόρων. Μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν ζητούσε από τον Οργανισμό Περιβάλλοντος να εμβαθύνει στην ε, έρευνα της αξιοπιστίας και της διαχείρισης επεξεργασίας των δεδομένων κατά την ανάλυση των συνεπειών των διαφόρων πολιτικών και την ε, ε, πρόταση συγκεκριμένων σεναρίων πολιτικών ανάλογα με τα πορίσματα των εκθέσεων. Βέβαια, ε, δεν ήταν αυτή δεν είχε αυτό τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί υπήρχαν κάποιοι σκεπτικιστές εκεί. Μερικοί ήταν κατά οποιασδήποτε ανάλυση των πολιτικών η ανάλυση της εφαρμογής των πολιτικών από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Αλλά σήμερα χαιρόμαστε ιδιαίτερος γιατί φαίνεται ότι όλοι είναι ικανοποιημένοι από την πορεία που πήραν οι εργασίες στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Θεωρώ ότι αυτή η σταθερή ε, και ε, ισχυρή ενθάρρυνση του οργανισμού να στηρίξει τον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις παγκόσμιες συζητήσεις για το περιβάλλον και στα θέματα αηφόρου ανάπτυξης, πράσινης καινοτομίας, κυκλικής οικονομίας, φυσικού κεφαλαίου. Όλα αυτά, όπως προέκυψε και από τη συζήτηση, οδηγούν την, τον οργανισμό και το έργο του προς τη σωστή κατεύθυνση, ακολουθώντας φυσικά τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις καθοδηγήσεις. Και μάλιστα η μέχρι τώρα υποστήριξη ενισχύθηκε και με την παρουσίαση αυτής της έκθεσης και την ανάλυση των ε, μεγατάσεων ε, και το συμπέρασμα ότι οι περισσότερες προκλήσεις μας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα. Σε ό,τι αφορά το θέμα της αξιοπιστίας και της διαφάνειας των δεδομένων. Και από αυτήν την άποψη η έκθεση είναι καινοτόμα. Γιατί επιτρέπει εύκολη πρόσβαση όλων των πολιτών ε, στις στις πληροφορίες αυτές και σε ε, ακατέργαστα μερικές φορές ακόμη στοιχεία. Ε, μπορεί ο καθένας λοιπόν να έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά και ακόμη να αμφισβητήσει τις ερμηνείες που δίνει ο οργανισμός περιβάλλοντος. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος λοιπόν γιατί έγιναν, εισακούστηκαν οι προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέλος, ήθελα να πω ότι ε, οι αποτελεσματικές λύσεις με βάση συστηματικές και περιεκτικές ε, προσεγγίσεις προϋποθέτουν μία εμπεριστατωμένη και μακρόπνοη πολιτική που θα πρέπει να στηρίζεται σε όλα τα επίπεδα. Και θα πρέπει και η Επιτροπή σας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του να διδραματίσουν το ρόλο τους και σε συνεργασία με άλλα κοινοτικά θεσμικά όργανα να διατρανούν την ανάγκη της εφαρμογή της διαφάνειας και της κοινή λογική στη χάραξη και εφαρμογή των πολιτικών και της λήψης αποφάσεων. Και από αυτή την άποψη έχουμε την αίσθηση ότι στον οργανισμό περιβάλλοντος η ρεαλιστική προσέγγιση που μπορεί μερικές φορές να είναι απεσιόδοξη δίνει, φέρνει ταυτόχρονα και προσθέτει τα απαραίτητα στοιχεία για την χάραξη και εφαρμογή πολιτικών με πολύ αισιόδοξο τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Και τώρα, θέλετε το λόγο. Να προσθέσω και εγώ κάτι. Να ευχαριστήσω στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Τα τελευταία αυτά τρία χρόνια ήταν μια εξαιρετική εμπειρία και είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε και άλλη μια τριετή περίοδο. Θα ήθελα να αναφέρω ένα πράγμα. Αυτό είναι η αντίδραση και η ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας αυτής σε όλα μας τα σχόλια ήδη από τις ε, πρώτες φάσεις της Ευρωπαϊκής Έκθεσης. Μπορώ να πω πως ε, πολλά από τα σχόλια μας ε, ελήφθησαν υπόψη και νομίζω πως αντιχούν και αυτά τα οποία ακούστηκαν εδώ μέσα. Από οποία αφορά την ε, αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, την κυκλική οικονομία, αλλά και την οικονομική λογική μιας ε, στιβαρής ε, περιβαλλοντικής πολιτικής. Και ακούσατε πράγματι και το που θα εστιάσει το μέλλον η Ευρωπαϊκή Έκθεση Περιβάλλοντος. Είμαι ευγνώμων για όλα αυτά και για το ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος υιοθέτησε κάποια από τα σχόλια που είχαμε κάνει και εγκρίνει ως δικά της ε, σχόλια. Πρόκειται λοιπόν για πάρα πολύ καλή και ανοιχτή συνεργασία και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Και τώρα θα δώσω τον λόγο στον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Μπράινινγκς για να δώσει τις απαντήσεις του, αλλά πρέπει να περιοριστείτε σε 12 λεπτά. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και στις 94 ερωτήσεις που έγιναν. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ για τα θετικά σας ε, σχόλια και θα ήθελα να αναφέρω δύο ζητήματα που έθιξαν οι βουλευτές. Πρώτα απ' όλα η διαφάνεια και η χνηλασιμότητα των δεδομένων της έκθεσης γιατί εστιάστηκα στα μηνύματα της πολιτικής, αλλά βεβαίως ε, βασίζονται στην πολύ καλή παρακολούθηση του περιβάλλοντος της Ευρώπης ε, στα κράτη-μέλη. Και μπορείτε πραγματικά να μπείτε σε οποιοδήποτε θέμα, να πατήσετε σε ένα χάρτη, θα ανοίξει ένα κουτί με τα βασικά δεδομένα και μπορείτε να τα δείτε. Οπότε η διαφάνεια, η εχνηλασιμότητα είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς και νομίζω πως είμαστε πρώτοι στον κόσμο. Δεν θα βρείτε ε, πουθενά αλλού 39 χώρες να μοιράζονται τα βασικά δεδομένα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό από πλευράς ε, διαφάνειας. Ε, επίσης να πω πως είναι μια έκθεση που προέκυψε από το δίκτυό μας και αυτό βεβαίως περιλαμβάνει και το Κοινοβούλιο. Στην συνθετική αυτή έκθεση λάβουν πάνω από 1500 σχόλια. Πολύ δουλειά λοιπόν που έπρεπε να γίνει, αλλά νομίζω πως έτσι αυξάνεται και η νομοποίηση της δουλειάς μας. Μία από τις ερωτήσεις, προτάσεις ήταν να παρουσιαστεί αυτή η έκθεση στις χώρες και στους ε, αρχηγούς κρατών. Θα έλεγα πως κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο έργο προς αυτή την κατεύθυνση με πάνω από 25 χώρες Οπότε θα έλεγα πως ε, μπορούμε να πάμε να παρουσιάσουμε την έκθεση, να πούμε ποια είναι τα σημαντικά για αυτή την χώρα και θα έλεγα πως ε, πραγματικά ε, θα μπορέσουμε έτσι να δώσουμε κάποιο βάρος. Μετά κάποια πιο λεπτομερή ζητήματα. Το θέμα της εφαρμογής, την όλη αυτή συζήτηση για το αν δεν χρειαζόμαστε πολιτική, αν χρειάζεται μια επιπρόσθετη πολιτική ή αν πρέπει να εστιάσουμε στην εφαρμογή. Δεν είναι μία η απάντηση σε κάποια άλλα ζητήματα. Είναι σαφές πως η πλήρης εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας είναι ένα τεράστιο βήμα πρόοδο. Αυτό ισχύει για τη βιοπικιλότητα, την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, όπου θα έχουμε ένα καλό καθεστώς ε, για το 50% μέχρι το 2015. Επίσης για τα απόβλητα το ίδιο ισχύει. Κάποιες ερωτήσεις τώρα αφορούσαν γενικά θα έλεγα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο όταν μιλάμε για την νομοθεσία μας. Να αναφερθώ σε κάποια πράγματα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα υπάρχει αυτή η υπόθεση ότι δηλαδή οι εταιρείες θα πάνε στη περιοχή εκείνη όπου είναι πιο χαλαρή η περιβαλλοντική νομοθεσία. Πρέπει να είμαι σαφής. Ελάχιστα πράγματα δείχνουν κάτι τέτοιο. Όταν οι εταιρείε μετακομίζουν, ο λόγος είναι το κόστος της εργασίας, του κοινωνικού συστήματος, για λόγους διείσδησης αγοράς και σε κάποιες περιπτώσεις το κόστος της ενέργειας. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μας λέει πως αυτό γίνεται για λόγους περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι ελάχιστο μέρος του κόστους ε, των επιχειρήσεων και οι περισσότερες μεγάλες εταιρείε έχουν δικούς τους κανόνες που εφαρμόζουν ε, οπουδήποτε δραστηριοποιούνται. Δεύτερον, αν δούμε το κόστος ε, της ενέργειας δεν είναι το κόστος ε, της ε, κιλοβατόρας που έχει σημασία, αλλά το κόστος αναμονάδα προϊόντος. Ε, και υπ' αυτή την έννοια έχει πολύ αποτελεσματική οικονομία και βιομηχανία η Ευρώπη σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Οπότε πρέπει να δούμε την παραγωγικότητα της ενέργειας και των πόρων και με έτσι το βλέπουμε διαφορετικά βεβαίως. Σας δώσω ένα χοντρικό νούμερο. Η αμερικανική οικονομία ε, ε, έχει διπλάσια ένταση ενέργειας αναπαραγόμενη μονάδα σε σχέση με μας. Οπότε έχουμε ένα πλέον έκτημα αν παράγουμε με τρόπο πιο αποτελεσματικό. Για την κυκλική οικονομία τώρα και τις πράσινες θέσεις εργασίας ε, βεβαίως είναι απολύτως σαφές και σημαντικό πως όταν η πράσινη οικονομία ή η κυκλική οικονομία όπως έρθει αυτό το πακέτο θα πρέπει να εστιάσει στην αποτελεσματική χρήση των πόρων ε, με έναν τρόπο προς τα ανάντη. Και έτσι ερχόμαστε στο πακέτο περί αποβλήτων. Και μιλήσατε για μια ιεραρχία απορριμμάτων Βεβαίως μιλάμε και για τον σχεδιασμό αλλά και για ζητήματα ποιότητας προϊόντων αυτή την λεγόμενη πρόγραμμα, τα, το, κάποια προϊόντα προγραμματίζονται να είναι παροχημένα και μετά από κάνα δύο χρόνια παραδείγματο χάρη δεν υπάρχουν αναβαθμίσεις ή δεν μπορούν να επισκευαστούν ή δεν υπάρχουν ανταλλακτικά Όλα αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά όταν, έχει κάποιος, ε, όταν θέλει κάποιος να κάνει την οικονομία πιο κυκλική. Κάτι άλλο το οποίο αναφέραμε στην έκθεση είναι η σημασία των επιχειρηματικών μοντέλων ε, από την ιδιοκτησία να περάσουμε στις υπηρεσίες. Τώρα σε κάποια μέρη της Ευρώπης μισθώνει κανείς και χημικές ουσίες, δηλαδή είναι θέματα όχι μόνο τεχνολογίας αλλά και το πώς προσεγγίζει τα υλικά και τα απορρίμματα. Όταν μιλάμε για τις πάρα πολύ μεγάλες διαφορές ε, που αναφέρθηκαν στα απορρίμματα. Δεν είναι μόνο εκεί οι διαφορές, ε, το βλέπει κανείς παντού. Οι διαφορές μεταξύ των κρατών είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και η Ευρώπη νομίζω έχει παίξει σε δύο επίπεδα. Έχουμε αφενός χρονικούς ορίζοντες και δίνουμε σε κάποια κράτη-μέλη και σε κάποιες διαδικασίες περισσότερο χρόνο και από την άλλη έχουμε διαφορετικούς στόχους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε άλλες πολιτικές. Πρέπει να λάβουμε υπόψη βεβαίω το πλαίσιο των χωρών, αλλά ο γενικός στόχος θα πρέπει να είναι να πηγαίνουν τα πράγματα στη σωστή κατεύθυνση. Είναι ένα θέμα ισορροπίας μεταξύ γενικών ευρωπαϊκών φιλοδοξιών και βεβαίως να φροντίσουμε όλα τα πρόβατα να ακολουθούν τον τζοπάνι. Γιατί αν θεωρεί κανείς προς, πως είναι ηγέτης αλλά δεν τον ακολουθεί κανείς δεν είναι ηγέτης, απλά πηγαίνει βόλτα. Και όσον αφορά τις ε, κοινωνικές επιστήμες και τον ρόλο των αξιών κτλ. Να πω το εξής. Ε, εμφανίστηκε ένα άρθρο όταν ανέλαβα καθήκοντα και έλεγε μα ένας κοινωνικός επιστήμονας τώρα αναλαμβάνει με μια επιστημονική υπηρεσία. Υπάρχει μια ένταση λοιπόν μεταξύ της πολιτικο-οικονομικής διάστασης και της επιστημονικής. θα έχουμε ενισχύσει αυτά. Ε, κάναμε και μια έκθεση για την ε, κατανάλωση και τονίζουμε και τον ρόλο της ε, πληροφόρησης ε, και τον ΜΜΕ για να αλλάξουν οι συνθήκες Όταν μιλάμε για την γαλάζια οικονομία... και το ίδιο ισχύει και για την πράσινη οικονομία. Αν δεν υπάρχει ένα ισχυρό θαλάσσιο στοιχείο δεν μπορεί να οικοδομήσει κανείς ε, μια βιώσιμη οικονομία υπηρεσιών και ξέρουμε πως έχουμε ε, ελλείμματα γνώσης ε, όταν μιλάμε για το θαλάσσιο περιβάλλον σε σχέση με το χερσαίο για την Ατούρα 2000 και τον ρόλο κοινωνικο-οικονομικών πτυχών ε, σε σχέση με το περιβάλλον, οι αγρότες, ο ρόλος των ανθρωπίνων όντων ε, και η αγροτική ανάπτυξη και οι δουλειές. Είναι σαφές πως ε, σε πολλές εκθέσεις ζητάμε μια ολοκληρωμένη πολιτική όταν μιλάμε για περιβαλλοντικούς ε, και κλιματικούς στόχους στην κυνηγιορική πολιτική, η οποία βεβαίως σαφώς έχει επίκεντρο τους αγρότες και τη γεωργική παραγωγή. Είναι σαφές ε, πως ε, η οδηγία των αζωτούχων ή Natura 2000 των υδάτων έχουν διαφορετική κατεύθυνση και πρέπει να βρούμε κάποια κοινά στοιχεία και ωφέλη αυτή τη γραμμή ακολουθούμε εδώ και καιρό και έχουμε, το έχουμε τονίσει αυτό και στην έκθεση για τη γεωργία και τη φύση και θα καταθέσουμε μια νέα έκθεση. Νομίζω λοιπόν πως έχετε δει και όταν μιλάτε για ισορροπία χωρίς ποτέ να ξεχνάμε την κατεύθυνση της βελτίωσης του φυσικού κεφαλαίου. Εδώ πρέπει να είμαι σαφής, έτσι. Λοιπόν, για το έδαφος. Δεν χαράζουμε εμείς ε, την πολιτική, δεν θα πω εγώ ότι χρειαζόμαστε οδηγία για το έδαφος, αλλά είναι σαφές από τις εκθέσεις μας πως ε, το έδαφος ε, παίζει σημαντικό ρόλο στα οικοσυστήματα και υποτιμημένο. Καλλιεργούμε τις τροφές μας, παίζει ρόλο στον κύκλο του νερού, του άνθρακα επίσης, οπότε η εστίαση συμπιότητα του εδάφους από μια οικοσυστημική σκοπιά είναι πολύ σημαντική τώρα. Αν θα πάμε σε νέα κατεύθυνση όχι, αυτό επαφιέται στη σοφία αυτών που κάνουν την, και χαράζουν την πολιτική. Για την ανταγωνιστικότητα της πράσινης οικονομίας και για συγκεκριμένα παραδείγματα τώρα αυτό σαφώς ισχύει στην αποτελεσματική χρήση της ενέργειας που έχουμε πρώτες στον κόσμο εταιρείε, ανανεώσιμες πηγές, ε, ο τομέας των χημικών με πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση πηγαίνει σε μια πιο βιολογική χημεία αλλά και σε συστήματα αστικών μεταφορών ή αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη έχει κάνει πάρα πολλές καινοτομίες, ε, ανακύκλωση το βλέπετε αυτό, είναι κομμάτι της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας όταν μιλάμε για ανταγωνιστικότητα. Μετά για την εμπλοκή των πολιτών, ε, αναφέρθηκε το Noise Watch ε, και τα λοιπά. Πράγματι η εμπλοκή των πολιτών είναι σημαντική όταν μιλάμε για να οικοδομήσουμε μια βάση περιβαλλοντικών πολιτικών. Το εάν θέλουμε τώρα να αναπτύξουμε και άλλες τέτοιες εφαρμογές έδωσα μία απάντηση που ε, δεν μου άρεσε. Δεν θέλω να κλαίγομαι τώρα για τους πόρους και τα σχετικά αλλά ε, είμαστε εντός των ορίων του προπολογισμού και κάθε χρόνο χάνουμε προσωπικό. Οι πόροι μας λοιπόν είναι πολύ περιορισμένοι. και ήμασταν ε, ιδρυτικό μέλος ε, του δικτύου πολιτών επιστημόνων και παίξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη συλλογή και διάθεση δεδομένων εντελώς δωρεάν. Αλλά είμαστε πάρα πολύ περιορισμένοι όσον αφορά τους πόρους. Μετά για την χρηματοδότηση τελειώνω Υπάρχει πολύ δημόσιο χρήμα στην οικονομία ήδη. Βασικό ερώτημα είναι ποια είναι η κατεύθυνση, η μακροοικονομική και μακροκοινωνική κατεύθυνση στην οποία κατευθύνονται αυτά τα χρήματα. Και πράγματι αυτό ισχύει για τις στρατηγικές επενδύσεις όπου τρεις από τις πέντε προϋποθέσεις ε, σχετίζονται με αυτό. Ε, χρήση πόρων, φυσικό κεφάλαιο, μείωση του άνθρακα καινοτομία. Οπότε υπάρχουν αυτά. Στα φορολογικά συστήματα πάρα πολύ δουλειά έχει γίνει. Για τους ε, φόρους επίσης αφήσει σύσταση και στο εξάμεινο, επιδοτήσεις ε, βλαπτικές προς το περιβάλλον, περιλαμβάνονται. Είναι θέμα λοιπόν πολιτικής κατεύθυνσης που πρέπει να δοθεί στα κονδύλια αυτά. δύο πραγματάκια ακόμα όταν μιλάμε για πόρους εκτός Ευρώπης, σπάνιες γιές και Αρκτική. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια έκθεση για την Αρκτική. Θα έχει τελειώσει μέχρι το τέλος του έτους για να στηρίξει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αρκτική. Είναι προφανές πως είναι ευαίσθητο το θέμα και η περιοχή αυτή του πλανήτη. Δεν μιλάω μόνο πολιτικά ευαίσθητη αλλά και περιβαλλοντικά. Υπάρχει ελάχιστη διακυβέρνηση, οπότε οι κανόνες είναι ε, ελάχιστοι και αν σκεφτεί κανείς κάποιον προϋπολογισμό άνθρακα, εάν θέμε να μείνουμε κάτω από τους δύο βαθμούς έχουμε περισσότερους πόρους από όσους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή. Το θέμα λοιπόν είναι πώς θα μεταφραστούν αυτά σε συγκεκριμένους κανόνες. Αυτός είναι ο ρόλος των πολιτικών. Όταν μιλάμε για το εμπόριο, τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, ε, εμείς ελάχιστο ρόλο έχουμε να παίξουμε, δεν έχουμε τους πόρους να μπούμε σε αυτή την κουβέντα, οπότε δεν έχουμε κάποιο ρόλο για την ώρα. Αυτό το οποίο κάναμε ήταν να κοιτάξουμε το εμπορικό ισοζύγιο και το πώς εξωτερικοποιείται το αποτύπωμά μας ε, συχνά μέσω εμπορικών κανόνων ε, για ενέργεια, πόρους, ε, χρήση γης και αυτό νομίζω μπορεί να συνεισφέρει στη συζήτηση, αλλά λίγα πράγματα κάνουμε. Με συγχωρείτε αν μακρηγόρησα, υπήρχαν πολλά ζητήματα, ελπίζω να μην απογοήτευσα κάποιον αν δεν απάντησα στην ερώτησή του. Για περισσότερες απαντήσεις ελάτε σε επαφή μαζί μας. Πάντα απαντάμε σύντομα με τις πληροφορίες που ζητάτε. Ελάτε λοιπόν σε επαφή μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα περνάμε αμέσως στο επόμενο θέμα γιατί έχουμε καθυστερήσει. Το επόμενο σημείο προβλέπει την εξέταση της γνωμοδότησης, του σχεδίου γνωμοδότησης με θέμα τις φαρμακούχες ζωοτροφές. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον εισηγητή, στον συντάκτη γνωμοδότη, στον κύριο Λίντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την δυνατότητα που μου δίνετε να παρουσιάσω τη γνωμοδότησή μου για τις φαρμακούχες ε, ζωοτροφές. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κατατάξουμε την υπόθεση αυτή. Πρόκειται για ένα μέρος του συνολικού πακέτου φαρμακούχων ε, ζωοτροφών. Αφενός υπάρχει ο κανονισμός για τα ε, ζωικά φάρμακα της κυρίας Γκροστέτ. Η δεύτερη είναι τα φάρμακα στις ε, ζωοτροφές ε, που απασχολούν βεβαίως την Επιτροπή Γεωργίας και το τρίτο κομμάτι είναι μια πρόταση κανονισμού για την σύσταση μιας σχετικής ευρωπαϊκής υπηρεσίας ως εισηγητής είναι για μένα σημαντικό να ε, μπορέσουμε να συνεννοηθούμε έτσι ώστε στο τέλος να έχουμε ένα κείμενο το οποίο θα έχει μια συνοχή. Πρέπει να υπάρχει και νομική ασφάλεια για τους χρήστες και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην υπάρχουν διάφορες ε, διαιρέσεις ε, για τα ε, φαρμακούχες ε, ζωοτροφές ε, και τον σχετικό κανονισμό. Θα πρέπει να δούμε γενικώ τι γίνεται με τις αντιμικροβιακές δραστικές ουσίες και να έχουμε και σαφείς ορισμούς για τις διάφορες μόρφες θεραπείας, την θεραπευτική, την μεταφυλακτική κλπ και την προληπτική. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Νομίζω πως τα χρονοδιαγράμματα συγκλίνουν. Και το ίδιο συμβαίνει και με την ε, προσέγγιση μας. Ε, χαιρετίζω την πρόταση της ε, Κομισιόν και νομίζω πως είναι σωστό εδώ πέρα να οδηγηθούμε σε μια εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά Νομίζω πως είμαστε σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο. Η επιλογή δε του κανονισμού ως νομικού μέσου είναι πάρα πολύ σημαντική. Η παλαιά οδηγία η οποία ήταν από το 1990 ε, νομίζω έχει φτάσει η στιγμή να αντικατασταθεί. Θα καταλήξουμε λοιπόν σε καλύτερη υγεία των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα λάβουμε υπόψη ε, και την υγεία ανθρώπων και ζώων. Και βεβαίως το ότι είναι συνδεδεμένες αυτές οι δύο πτυχές. Ποιο είναι το θέμα μας λοιπόν εδώ πέρα. οι φαρμακούχες ζωοτροφές ε, είναι ζωοτροφές οι οποίες περιέχουν ε, φαρμακευτικές ε, δραστικές ουσίες, συχνά και αντιβιωτικά. Δεν είναι έτοιμα φάρμακα τα οποία μπαίνουν μέσα στο νερό ή σκορπίζονται μέσα στην ζωοτροφή. Πρόκειται για ουσίες που χρησιμοποιούνται σε μεγάλα κοπάδια ζώων, πουλερικά ή και ψάρια ή χείρους. Βεβαίως οι διατάξεις αυτές θα ισχύσουν ε, και για τα κατοικίδια ζώα συγκεκριμένα. Λοιπόν, το θέμα είναι ποιος μπορεί να ε, χρησιμοποιήσει και να αναμίξει τις ουσίες αυτές, ε, συγκεκριμένα οι αγρότες δηλαδή. Το θέμα είναι μετά πώς γίνεται αυτό, το θέμα δηλαδή των οριακών τιμών και το θέμα της χρονικής διάρκειας της ε, χρήσης. Επιπλέον γίνεται διάκριση μεταξύ αντιμικροβιακών και μη δραστικών ουσιών. Ποιοι είναι οι στόχοι, ε, αυτονόητο βεβαίως ε, είναι πως ε, στόχος είναι το πρόβλημα της αυξανόμενης αντίστασης αντοχής στα αντιβιωτικά Δεν είναι μόνο αυτό όμως, είναι και το ζήτημα της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της διαθεσιμότητας των φαρμακών αυτών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προτείνω συγκεκριμένα τώρα τέσσερις τομείς που πρέπει να αλλάξει η πρόταση της Κομισιόν. Πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο ήδη αναφέρθηκε, οι σαφείς ορισμοί των αντιμικροβιακών δραστικών ουσιών, οι διαφορετικές μορφές χρήσης ε, και να πέρα να έρθω και σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους εισηγητές ε, στις υπόλοιπες ε, εκθέσεις για να καταλήξουμε σε μια ενιαία αντιμετώπιση και στις τρεις, στους τρεις μετά. Προτείνω, όπως είπα, μια προληπτική αντιμετώπιση, μια απαγόρευση της προληπτικής ε, αντιμετώπισης και βεβαίως ε, ενισχύουμε τον ρόλο των κτηνιάτρων ε, του βασικού δηλαδή υπεύθυνου στην όλη διαδικασία και η συνταγογράφηση των φαρμάκων αυτών θα γίνεται μετά από υποχρεωτική εξέταση και επίσκεψη και το θέμα είναι μετά βεβαίως πόσο επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται αυτά τα φάρμακα. Η Κομισιόν προτείνει 14 ε, ημέρες, εγώ το μείωσα στις 7 ημέρες γιατί η χρήση των αντιβιωτικών ε, ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται μετά τις 7 ημέρες. Για το θέμα τώρα της ε, μεταφοράς ε, προτείνω κάποιες ε, φιλόδοξες προσεγγίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά αντιλαμβάνομαι πως και η ΕΦΣΑ θα ε, κάνει μια επιστημονική αξιολόγηση κινδύνου για τις ε, συγκεκριμένες ειδικέ ε, και μη τιμές μεταφοράς. Αυτά από μένα. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την συνεργασία με τους σκιοδησηγητές. Αναμένουμε τροπολογίες μέχρι τις 24 Απριλίου και 17 Ιουνίου προβλέπεται η ε, ψήφιση της έκθεσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στη συζήτηση. Πρώτα στους και διησηγητές, ε, ο λόγος ο κ. Τζάνι. Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ε, θα ήθελα να επαναλάβω και να τονίσω όλους όσους παρακολουθούν στις συζητήσεις ότι μιλούμε για ένα νέο κανονισμό, μια νέα πρόταση κανονισμού η πρόταση ε, και οι τροπολογίες ε, ακολουθούν μία κατεύθυνση, ε, την εξασφάλιση της υγείας και των ανθρώπων και των ζώων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε και οι παρασκευαστές φαρμακούχων ζωοτροφών να μπορούν να χορηγούν τα προϊόντα αυτά, αλλά μόνο μετά από συνταγογράφηση από κτηνίατρο. Φυσικά θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές και στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπής, ως ήθιστε, αλλά θεωρώ ότι η γνωμοδότηση του κυρίου Λίνς είναι πολύ αξιόλογη και είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες ε, για αρκετά θέματα. Ήδη έχει γίνει η προεργασία και έχουμε συμφωνήσει σε πολλά θέματα στην πρώτη συνεδρίαση των σχεδόν εισηγητών. Για να αποφύγουμε επαναλήψεις, εγώ θα σταθώ σε τέσσερα σημεία. Θεωρώ ότι οι φαρμακούχες ζωοτροφές είναι πολύ σημαντικός τρόπος για τη χορήγηση φαρμάκων στα ζώα. Δεύτερο σημαντικό θέμα αφορά την υγεία. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού το θέμα της υγείας των ανθρώπων και των ζώων και να εξασφαλίσουμε την υγεία και των ανθρώπων και των ζώων. Τρίτον, ο ρόλος των κτηνιάτρων αναμφισβήτητος και αδιαφιλονίκητος ο ρόλος ε, των ε, κτηνιάτρων και επίσης ε, να εντοπίσουμε τα κτηνιατρικά θέματα και τις φάρμακα και τις δραστικές ουσίες. Και ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο θέμα στην οδηγία για τα κτηνιατρικά φάρμακα θα πρέπει να έχουμε μια σχετική ευθυγράμμιση των οδηγιών για να αποφεύγουμε τις επαναλήψεις. Πάντως η σχετική πρόταση θα πρέπει να δώσει ενάψματα για έρευνα σε φαρμακούχες ζωοτροφές. Είναι υπέρ αυτών των κινήτρων και η ομάδα των σοσιαλιστών και προσβλέπω στη συνέχιση της συζήτησης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκολσον από τους μεταρρυθμιστές συντηρητικούς. Ευχαριστώ. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους χορήγησης κτηνιατρικό φαρμάκων είναι οι φαρμακούχες ζωοτροφές. Ήταν πολύ χρήσιμη η συνεισφορά του στην καταπολέμηση επιζωτιών. Και 25 χρόνια μετά από την αρχική οδηγία χρειαζόμαστε πια νέα μέτρα, γιατί πρέπει να παρακολουθούμε την τεχνολογική πρόοδο και να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και για τους παραγωγούς και για τους ακτινοτρόφους. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή, το συντάκτη της γνωμοδότης για τη σημαντική του συνεισφορά. Συμφωνώ με πολλέ τροπολογίε του, για παράδειγμα της, ε, ε, τη συμπερίληψη και των ζώων που δεν προορίζονται για παρασκευή τροφίμων και επίσης θα πρέπει να κάνουμε κάτι με τα όρια τη μεταφορά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις τιμές μεταφοράς που προτείνει στο άρθρο 7 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. σαφώ καθορισμένα όρια και τιμές ίσως είναι καλά για την ασφάλεια δικαίου, αλλά το όριο του 1% για τις αντιμικροβιακές δραστικές ουσίες ε, ε, δεν είναι ευχριστή λύση, ούτε αναλογική με τους προτινόμενους κινδύνους. Αν θέλουμε να πετύχουμε αυτό το κατόφλι, θέλουμε τουλάχιστον ε, πιο μεγάλη μεταβατική περίοδο για την υλοποίηση του στόχου. Αλλιώς θα φέρουμε σε πολύ δύσκολη θέση τον κλάδο. Υπάρχουν όμως κάποιες τροπολογίες που δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Για παράδειγμα, η τροπολογία 14, πολύ φοβούμαι ότι θα έχει ανεπιθύμητες συνέπειες. Στο Ενωμένο Βασίλειο, από που και κατάγομαι, έχουμε αρκετούς ικανούς ανθρώπους που μπορούν να συνταγογραφήσουν τέτοια τέτοιε φαρμακούχε ζωτροφέ και που δεν είναι, δεν είναι όλοι κτηνίατροι, άρα δεν εμπίπτουν στην οδηγία για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Και ο περιορισμό τη συνταγογράφηση μόνο στου κτηνιάτρου ίσω ε, περιορίσει τι δυνατότητε που έχουν οι κτηνοτρόφοι και ουσιαστικά υπονομεύσει το ρόλο ανθρώπων που έχουν ε, ε, προσόντα και γνώσει για τέτοια συνταγογράφηση. Επίση, στο σημείο 17, για την αποφυγή της κατάχρησης ο αρμόδιος επίτροπος στην Επιτροπή Άγκρη είχε πει ότι θα πρέπει ότι ήταν υπέρ της απαγόρευσης της προληπτικής αγωγής, της προληπτικής χρήσης φαρμάκων. Εγώ δεν συμφωνώ. Συμφωνώ βέβαια ότι ε, οι φαρμακούχοι ζωοτροφές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ανάπτυξης των ζώων, αλλά το σημείο 17 κατά τη γνώμη είναι υπερβολικά περιοριστικό, γιατί μερικές φορές η προληπτική αγωγή διορθώνει ε, μερικά λάθη στη διαχείριση Και μερικές φορές, όπως ξέρουμε μάλλον, η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Δεν θα πρέπει λοιπόν να την απαγορεύουμε ε, ολοσχερό στην προληπτική αγωγή. Άλλωστε, μερικές φορές χρειάζεται ε, χρόνο για να δράσουν τα φάρμακα και μερικά αρχικά συμπτώματα μπορεί να είναι ε, συμπτώματα σημαντικής ε, Οπότε αν έχουμε ολοσχερή απαγόρευση προληπτικής αγωγής θα βρεθούμε μερικές φορές προτελεσμένο γεγονότο και θα χρειαστεί πολύ αργά πια, σε πολύ προχωρημένο στάδιο της νόσου, ε, να δώσουμε φαρμακευτική αγωγή. Πολύ ενδιαφέρουσα πάντως η γνωμοδότηση. Έχουμε κάποια προβλήματα, αλλά θα συνεργαστούμε με τον συντάκτη για να τα υπερκεράσουμε. Ευχαριστώ. Τώρα εξ των Πρασίνων ο κύριος Όσλιν. Είπα και στην προηγούμενη συζήτηση πως είμαι πολύ επικριτικός απέναντι στον κανονισμό γιατί δεν υπάρχουν στόχοι μείωσης σε σχέση με τον παλιό κανονισμό και ειδικά για τα αντιβιωτικά στις ζωοτροφές είμαι πάρα πολύ επικριτικός. Και δυστυχώς η Κομισιόν εδώ πέρα δεν είναι πολύ συνεπής ε, καθώς λέτε θέλει συνολικά να μειώσει τη χρήση αντιβιωτικών. Αυτό το οποίο προτείνει τώρα ο εισηγητής θα είναι καλό, αλλά βεβαίως θα θέλαμε μία βελτίωση. Έχουμε απαγόρευση της προληπτικής ε, χρήσης. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα εφαρμογής. Το δεύτερο, η, ε, η ελέγχου. Κοιτάξτε, κάποια είδη ζώων δεν γίνεται να α, ε, λάβουν φάρμακο παρά μόνο μέσω της ε, ζωοτροφής. Μα αν μιλάμε για μεγάλα ζώα όπως τα γουρούνια και λέμε ότι δεν μπορούμε να τους δώσουμε φάρμακο με άλλο τρόπο, πρέπει να δούμε συνολικά το σύστημα. Εγώ δεν σκοπεύω να μείνει η χρήση του ελέγχου έχει τώρα. Ε, η ενίσχυση του ρόλου των κτηνιάτρων, σωστή, αλλά οι κτηνίατροι σε κάποια συστήματα επωφελούνται από την χρήση κτηνιατρικών ε, φαρμάκων. Δεν θα πρέπει να έχουν συμφέρον να προωθούν τέτοια φάρμακα. Λοιπόν πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ αυτών που γράφουν την ε, συνταγή και αυτών που ε, χορηγούν μετά. Τώρα οι οριακές τιμές για τη μεταφορά είναι πάρα πολύ υψηλές, θα πρέπει να πέσουν ειδικά εάν σκεφτούμε πως ε, σε μικτές ε, μεταφορές από τη μία στην άλλη επιχείρηση υπάρχουν ε, προβλήματα, ειδικά αν σκεφτούμε πως σε μία εκμετάλλευση, παραδείγματο χάρη έχουμε γουρούνια και στην επόμενη μετά βοηδή. Τώρα για την προθεσμία 14 μέρες είναι πάρα πολλές, 7 μέρες να το δεχτούμε. Οπότε η έκθεση πάει προς σωστή κατεύθυνση. Το βασικό πρόβλημα για εμάς του πράσινους είναι όλη αυτή η προσέγγιση που είναι λάθη, λάθος. Και ε, στο πλαίσιο αυτό, εν πάση περιπτώσει, συμφωνούμε με τον εισηγητή πως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες για να περιορίσουμε ακόμη περισσότερο τη χρήση. Ο κύριος Πεντατσίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς ε, με μια πρώτη ανάγνωση είμαστε υπέρ της πρότασης ε, κανονισμού για τις ε, φαρμακούχε φαρμακούχες ζωοτροφές, κυρίως για τα θέματα που αφορούν την προστασία της ανθρώπινης υγείας, και ελπίζουμε τουλάχιστον σε αυτούς τους κανόνες να μεταφερθούν κάποια από τα μέτρα που έχουμε κάνει στις προτάσεις ε, πρωτοβουλίας για την ε, μικροβιακή εντοχή και την ασφάλεια των ασθενών. Η θέση μας λοιπόν είναι γνωστή. Ε, σε γενικές γραμμές θα προτιμούσε και για τα ζώα όπως και για τους ανθρώπους οι θεραπείες να είναι εξο, εξατομικευμένες και να μην είναι ε, συνολικές. Γι' αυτό και είμαστε υπέρ μιας προσέγγισης η οποία στόχο έχει όσο το δυνατόν περισσότερη μίεση αν όχι και απαγόρευση της προληπτικής χρήσης. η χρήση ε, αντιμικροβιακών στοιχείων θα πρέπει να ε, μειωθεί στο ελάχιστο και θα πρέπει τουλάχιστον να καθορίσουμε ένα στόχο μείωσης, ένα δίκτυο ο οποίος θα είναι μετρήσιμος για τη χρήση αντιβιωτικών ε, στις ζωοτροφές. Επαναλαμβάνω όμως η απαγόρευση των φαρμακούχων ζωοτροφών ως ε, ενίσχυση της ανάπτυξης και θα πρέπει ίσως να υπάρχουν και πιο αυστηρά μέτρα και πιο αυστηρές κυρώσεις για όσους τα χρησιμοποιούν. Επίσης ε, χρήση αντιβιωτικών για να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε ελλείψεις σε υγειονομικά ζητήματα στους χώρους όπου ζουν τα ζώα. Ε, οι κτηνίατροι θα πρέπει να είναι οι μόνοι οι οποίοι θα συνταγογραφούν και θα χορηγούν τέτοια φάρμακα εάν επιτρέψουμε κάτι άλλο, ε, σημαίνει ότι επιτρέπουμε να υπάρχει κενό. Ε, βέβαια, οι κτηνίατροι δεν θα πρέπει να συνταγογραφούν και να πολλούν τα αντιβιωτικά. Ε, στις ζωοτροφές θα πρέπει να απογορεύεται να αποφεύγεται η χρήση ε, συγκεκριμένων ε, ε, ουσιών. Όσον αφορά τη μεταφορά, θεωρώ ότι το 3% στα κατάλοιπα φαρμάκων θα μπορούσε ίσως να μειωθεί κι άλλο. Και όσον αφορά και το χρόνο συνταγογράφησης των αντιβιωτικών, συμφωνώ με τον συντάκτη ότι θα μπορούσαμε να είμαστε στη μία εβδομάδα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ανάγκη παρακολούθησης για το πόσες φορές επαναλαμβάνονται αυτές οι συνταγές, για να αποφύγουμε να μην υπάρχουν ανομαλίες στις ε, συνταγές ή να έχουμε επαναλαμβανόμενες ε, συνταγές. Ευχαριστώ και τώρα έχουμε 10 λεπτά για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Ε, πέντε άτομα έχουν ζητήσει το λόγο και πρέπει να αφήσουμε και χρόνο στην Κομισιόν. 1,5 λεπτό λοιπόν για κάθε ομιλητή. Θα προσπαθήσουμε να περιορίσουμε το χρόνο. Η κυρία Γκροστέτ. Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Καταρχάς να συγχαρώ το συνάδελφο τον κύριο Λίντς ε, για την εξαιρετική του δουλειά. Το κείμενο αυτό βασίζεται σε μεγάλο βαθμό με τον κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα και υπήρχε πολύ καλή συνεργασία. Προσπαθούμε να ενερμονίσουμε τις συνθήκες πορείε διάθεση στην αγορά και χρήση των φαρμακούχων ζωοτροφών για να είναι αποτελεσματικές, να είναι ασφαλείς για τη δημόσια υγεία και όλα αυτά συνδέονται φυσικά και με την υγεία των ζώων. Το βασικό ζήτημα και για τα δύο κείμενα είναι η αντιμικροβιακή εντοχή. Ε, πράγματι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτό το ε, θέμα το οποίο αποτελεί ε, λέλαπα για την δημόσια υγεία και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτή τη χρήση των όρων προφυλακτικών, ε, μεταφυλακτικών και ε, το, στις τροπολογίες 9 και 11. Εμείς είμαστε υπέρ και θα μπορούσα να δεχτώ και αυτούς τους ορισμούς και, και στην έκθεσή μου. Η προφυλακτική χορήγηση, η προληπτική συγγνώμη χορήγηση φαρμάκων και η απαγόρευση είναι κάτι το οποίο υποστηρίζω απόλυτα και θα το συμπεριλάβω και εγώ στην εκθεσή μου όσον αφορά τη χρήση των αντιβιωτικών σε κτηνιατρικά φάρμακα. Θέλουμε να υπάρχει απόλυτη συνέπεια μεταξύ των δύο κειμένων. Άκουσα και τι είχαν να πούνε οι σκιώδεις και θεωρώ ότι θα πρέπει να πλαισιώσουμε καταλήλως το ρόλο των κτηνιάτρων, τι διαφορά υπάρχει μεταξύ συνταγογράφησης και χορήγησης των φαρμάκων. Στη χορήγηση θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα και εγώ στην έκθεσή μου υποστηρίζω επίσης την ίδια άποψη. Δεν ε, θέλω να μακρηγορήσω άλλο, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να ε, μπορέσουμε να έχουμε μια σύμπνοια και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Επομένως θεωρώ ότι είναι θετικό. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκούτελαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα Καταρχάς να πω ότι κάθε χρόνο 25.000 άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πεθαίνουν εξαιτίας της μικροβιακής εισαντοχής. Και περί αυτού πρόκειται και στην συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Πώς θα καταπολεμήσουμε τη μικροβιακή αντοχή. Εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν. Πιστεύω ότι οι φαρμακούχες ζωτροφές δεν είναι η μοναδική λύση, αρκεί να βελτιώσουμε την υγεία των ζώων και να προσέξουμε την ευημερία τους. Τότε θα χρειαστούμε πολύ λιγότερες φαρμακούχες ζωοτροφές. Υπάρχει το πρόβλημα του υπερπληθισμού των χείρων στα χειροστάσια. Τεράστιο πρόβλημα. Αν δεν είχαμε τέτοιο συνοστισμό στα χειροστάσια, ε, δεν θα χρειαζόταν να χορηγούμε τόσες ε, φαρμακούχες ζωοτροφές. Θα πρέπει λοιπόν ε, να αναθεωρήσουμε τις πρακτικές εκτροφής περισσότερο. Η κυρία Σιέρικ Πίρικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βλέπουμε εδώ πέρα πως στην Ολλανδία έχουμε στόχο την μείωση κατά 6% των αντιβιωτικών, αλλά πρέπει να παραμείνουν και υγιεί τα ζώα και οι άνθρωποι βεβαίως ε, και να συνεχιστεί και η παραγωγή τροφίμων. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γι' αυτό ανησυχώ λίγο για αυτά τα οποία διαβάζω εδώ πέρα στην ε, έκθεση σας. Οπότε, εντάξει, εμείς ε, δεχόμαστε τις δικές σας ευαισθησίες, αλλά πρέπει και εσείς να σεβαστείτε τις δικές μας. Τα είπε και ο κύριος Νίκολσον και όπως είπα και πριν παίζει και ο άνθρωπος κάποιο ρόλο. Έχω τώρα κάποιες ε, ερωτήσεις. Ε, μιλήσατε για αντικοκυδιακά στην ε, έκθεση αυτή και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της αλλαγής της οποίας προτείνετε. πώς ζυγίσατε αν θέλετε τις δύο πτυχές μιας αλλαγής πολιτικής. Σας ευχαριστώ κυρία Μίλλερ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και τον εισηγητή για την έκθεση και για το ότι υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί οι οποίοι θα ισχύσουν οι ίδιοι σε όλα τα κράτη-μέλη. Βεβαίως ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, ο ορισμός, το τι είναι έτοιμο φάρμακο και το τι είναι φάρμακο σε ζωοτροφές και το τι είναι φαρμακού χαζοτροφή θα ξεκαθαρίσει μόνο όταν έχουμε έναν κατάλογο προϊόντων. Θέλουμε και εμείς να μειώσουμε την αντοχή στα αντιβιωτικά και βεβαίως πρώτοι από όλου το θέλουν οι γεωργοί και πρέπει να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Παρ' όλα αυτά θεωρώ πως στον κανονισμό αυτό υπάρχουν κάποια ζητήματα επίμαχα Πώς θα γίνει ο έλεγχος, ε, θα πρέπει ο κάθε αγρότης ο οποίος αναμειγνύει φάρμακα στη ζωοτροφή να είναι πιστοποιημένες, αυτό είναι το ερώτημα. Και αν ναι, θα ελέγχει μετά στα κράτη-μέλη. Εγώ γνωρίζω από την περιοχή μου πως για ολόκληρη την Βαβαρία υπάρχουν μόνο εννέα ελεγκτές ζωοτροφών. Αν είναι τώρα να πιστοποιηθεί κάθε αγροτική εκμετάλλευση, θα υπάρξουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες για να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ, Πιλάρα Ευχαριστώ. Καταρχήν να συγχαρώ το συντάκτη της γνωμοδότησης και να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η πρότασή της ε, μου φαίνεται καλή. Όπως είπε και η κυρία Γκροστέτ, ο κανονισμός αυτός συνδέεται άμεσα με τον αντίστοιχο κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε συνεπείς και να ε, προσέξουμε να μην υπάρχουν επικαλύψεις. Η τροπολογία 3 που λέει δεν επιτρέπεται η προληπτική αγωγή, η προληπτική χρήση, ενώ ο κανονισμός ε, για τα κτηνιατρικά φάρμακα δεν προβλέπει τέτοια απαγόρευση. Οπότε, βέβαια η κυρία Γκροσέτη μας είπε ότι θα αλλάξει. Πάντως, αν γίνει απαγόρευση θα πρέπει να γίνει στον άλλο κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα και όχι εδώ. Επίσης πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να μπορούμε να προσφεύγουμε στην προληπτική αγωγή μετά από σύσταση κτηνιάτρου. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 5 που μιλά για το σημείο εφαρμογή. Νομίζω ότι είναι σαφέστερη η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την τροπολογία ε, του Σε ό,τι αφορά τη μικροβιακή εντοχή, την προληπτική αγωγή και τα υπαλληλικά, οι τροπολογίες 8, 9, 10 και 11 με τους ορισμούς, αυτό, αυτές περισσότερο αφορούν τον άλλον κανονισμό. Θα πρέπει όμως, ε, αν είναι ίδιοι ορισμοί, εντάξει, απλώς το επαναλαμβάνουμε, αλλά να μην απάδουν. Σε ό,τι αφορά τον ε, Τη συνταγογράφηση θα πρέπει να δίνεται από κτηνίατρο. Και επίσης ε, να δούμε τι είναι η ε, προφύλαξη ρουτίνας, γιατί σε θεραπείες κατά παραστοκτόνων δεν μπορούμε να απαγορεύουμε προφυλακτική αγωγή. Αυτό εξαρτάται από τον ε, αρμόδιο που θα προβεί στη συνταγογράφηση. Ευχαριστώ να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Πογγελίνη, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τα σχόλιά της. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κυρίως ευχαριστώ τον συντάκτη της γνωμοδότησης και την Επιτροπή σας για το έγγραφο το οποίο μας υποβάλλατε. Προφανώς και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το έγγραφο αυτό και να πω ότι είμαστε και ικανοποιημένοι για αυτές τις πρώτες ε, αντιδράσεις διότι σε γενικές γραμμές οδεύουν ε, προς την ίδια κατεύθυνση και την ίδια προσέγγιση που θελήσαμε εμείς να ακολουθήσουμε ε, στην αρχική μας πρόταση. Υπό την έννοια ότι ένας από τους στόχους που θέλαμε να θέσουμε ήταν η ρύθμιση της χρήσης των φαρμακούχων ε, μέσω, των φαρμάκων συγγνώμη, μέσω της ε, χορήγησης ζωοτροφών και ως μέσο ε, ελέγχου της μικροβιακής αντοχής. Θεωρώ ότι ο στόχος λοιπόν είναι κοινό και αυτό είναι σαφές και δεν θα θέλαμε να παρεκκλίνουμε από αυτό το στόχο. Ε, λαμβάνοντας υπόψη, όπως σας είχα πει και όταν παρουσιάσαμε την ε, πρόταση στην Επιτροπή Γεωργίας, το θέμα της υγείας και της ευημερίας των ζώων μας ε, ε, με βάση φυσικά και την ανθρώπινη υγεία και τη δημόσια υγεία. Θεωρώ λοιπόν ότι οι στόχοι είναι αυτοί και επομένω το μέσο θα πρέπει να είναι ένα μέσο ε, αντίστοιχο αυτού που σας έχουμε προτείνει. Διότι δεν θα πρέπει να λησμονούμε βεβαίως ότι φέρπουν και οικονομικοί λόγοι για όλες τις καταστάσεις εκτροφής ε, και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτές τις πτυχές. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν, διότι θεωρώ ότι όσον αφορά την τοποθέτησή σας ε, είναι ε, η ίδια με τη δική μας και γι' αυτό και είμαστε ανοιχτοί και στις προτάσεις που μας έχετε κάνει. Τώρα, να περάσω λίγο στο ε, θέμα συζήτησης και τις ερωτήσεις που, που ετέθησαν. Σας επαναλαμβάνω ότι εμείς δεν έχουμε ε, πρόβλημα. Μπορούμε για παράδειγμα να επεκτείνουμε τη χρήση των φαρμακούχων ε, ε, ζωοτροφών και των ενδείξεων όχι μόνο στα ζώα ε, τα οποία παράγονται για ε, τρόφιμα ανθρώπινης χρήσης, αλλά και, και στα ζώα συντροφιάς, ε, τα οποία δεν αποτελούν βέβαια κεντρικό θέμα, αλλά και στη συγκεκριμένη κατηγορία ζώων υπάρχουν λόγοι υγείας και ευημερίας που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ε, λαμβάνοντας δε υπόψη ότι τα ζώα συντροφιάς ζουν όλο ένα και περισσότερο μαζί μας και επομένως η επέκταση των κανόνων αυτών και σε αυτούς σίγουρα είναι η πλέον κατάλληλη. Δεν θα πρέπει λοιπόν να αποκλείουμε και αυτό το ενδεχόμενο. Είδα ότι υπάρχει και κάποιο ενδιαφέρον ε, για τους ορισμούς. Εμείς συμφωνούμε ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν οι ορισμοί. Κάποιοι πρότειναν ε, ότι καλύτερο θα ήταν να διευκρινιστούν στον άλλο κανονισμό, ε, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο κανονισμοί, αναφέρομαι στον κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα και ο συγκεκριμένο κανονισμός, ε, έχουν άμεση σχέση, ε, εμείς ρυθμίζουμε ουσιαστικά ένα τμήμα των ε, ε, κτηνιατρικών φαρμάκων. Ε, θεωρώ ότι θα ήταν εξαιρετική ιδέα. Δεν... Είμαστε αντίθετοι στη συγκεκριμένη προσέγγιση, ούτε σε αυτή την περίπτωση. γιατί νομίζω ότι διευκολύνει λίγο τη δουλειά όλων μας. Ιστορικά, γιατί μπορούμε πλέον να μιλάμε για ιστορία, η οδηγία είναι 30 χρονών. Είμαστε πλέον ε, στα επίπεδα της ιστορίας. Ε, είχαμε κάποια προϊόντα τα οποία είχαν ε, ε, έγκριση και μπορούν να χρησιμοποιούνται στις φαρμακούχες ζωοτροφές και θέλουμε να συνεχίσει αυτή η διαδικασία και στο μέλλον. Ε, διότι και σε αυτή την περίπτωση σίγουρα ε, δεν θα θέλαμε προϊόντα τα οποία προορίζονται για να χρησιμοποιούνται και να διαλύονται σε πόσιμο νερό ή θα ε, ε, διαλύονται στην επιφάνεια των ζωοτροφών. Συγγνώμη, αν θέλετε να συνεχίσετε, θα πρέπει να συνεχίσετε στα αγγλικά, διότι θα σταματήσει η διερμηνία. Thank you. <laughs> no, I, I try to finish because apparently it's quite late.